Εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Δύο Φύλων σας καλωσορίζω σε ένα απόγευμα που ελπίζω να είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε δημόσια ακρόαση για το θέμα «Η γυναίκα σε διευθυντικά θέσεις». Εδώ θα γίνει ένας πρώτος γύρος συζητήσεων, ένα πρώτο πάνελ που θα αποτελέσει και το πρώτο τμήμα. Και το δεύτερο, το δεύτερο θα έχει ως θέμα τα πολιτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ισότητα ανδρών και γυναικών. Κατά τη δημόσια αυτή ακρόαση θα αναφερθούμε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας της δικής μας Επιτροπής και όπως ξέρετε η δημόσια αυτή ακρόαση αποτελεί τμήμα της γενικότερης ανάλυσης που αφορά αυτό το θέμα της έκθεσης. Καλωσορίζω λοιπόν μεταξύ των ε, όλους τους ομιλητές ιδιαίτερα δε καλωσορίζω την κυρία Κράτσα που είναι η εισηγήτριά μας στην οποία θα δώσω σε λίγο και το λόγο. Όπως ξέρετε η κυρία Κράτσα είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία της. Είναι επίσης συγγήτρια για την πρωτοβουλία αυτή που μας ενδιαφέρει όλες τόσο. Στην, θα αρχίσουμε ακούγοντας τα προκαταρκτικά της κυρίας Κράτσα και της δίνω μέσα στο λόγο. Ορίστε κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ε, είναι πολύ σημαντικό για μας ε, η διοργάνωση αυτής της ε, δημόσιας ακρόασης με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στα υψηλά επίπεδα των μεγάλων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή Γυναικών στην οποία βρίσκεστε σήμερα, για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της, έχει δώσει μεγάλες μάχες με επιτυχίες τόσο σε θέματα πρόθεσης της νομοθεσίας, όσο και σε θέματα ε, υιοθέτησης στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την πρόθεση των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε το θέμα της θέσης των γυναικών στην στα υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να ρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φως στους λόγους της ε, χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, στα εποπτικά συμβούλια, υπάρχουν διαφορετικοί όροι από χώρα σε χώρα, ε, των μεγάλων εταιριών. Ε, γνωρίζουμε λίγο πολύ τους λόγους που οι γυναίκες ε, δεν βρίσκονται σε θέσεις ευθύνη. Είναι το κοινωνικό σύστημα, είναι ο τρόπος διοργάνωσης των επιχειρήσεων, ο τρόπο, των επιχειρήσεων, οι ανάγκε που δημιουργούν επαγγελματικέ ε, ε, δραστηριότητε και υποχρεώσει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Είναι τα θέματα της ίδια της φιλοδοξία ε, των γυναικών, τα κοινωνικά στερεότυπα που βαραίνουν ακόμη. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι γενικό και παγκόσμιο. Υπάρχουν όμως χώρες που έχουν διαφορετικά επίπεδα, ε, καταφέρουν να έχουν διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής γυναικών, πιο ενθαρρυντικά ποσοστά ε, συμμετοχής γυναικών στα υψηλά επίπεδα. Ακόμη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά το θέμα αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο μιας εταιρική διακυβέρνησης στον κόσμο σήμερα. Ε, οι λόγοι είναι για την, μια καλύτερη δημοκρατία, ε, οι αποφάσεις είναι πιο αιτιολογημένες, πιο νομιμοποιημένες όταν παίρνονται από κοινού άνδρες και από γυναίκες. Αλλά αυτό θα είχε ένα αποτέλεσμα και στην οικονομία μας, διότι είναι αποδεδειγμένο ότι οι γυναίκες στα κέντρα που λαμβάνουν αποφάσεις όταν βρίσκονται, τότε οι αποφάσεις είναι πιο κοντά στην κοινωνία, είναι πιο ευέλικτες, λαμβάνουν υπόψη πιο πολύ τις παραμέτρους της, της πολύπλεκης παραγματικότητας. Η δημόσια κρόση που σήμερα διοργανώνουμε στο Κοινοβούλιο ε, έχει σκοπό λοιπόν να συγκεντρώσει τις απόψεις πολιτικών ε, ε, ή γυναικών εκπροσώπων φορέων με εμπειρία στα θέματα της προώθησης των γυναικών στα υψηλά επίπεδα αποφάσεων των μεγάλων εταιριών. Θα ανταλλάξουμε απόψεις μαζί, μεταξύ μας και θα είναι οπωσδήποτε χρήσιμες για να αξιολογήσουμε αυτά που ήδη έχουν συμβεί, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν χώρες που έχουν μια θετική εμπειρία να μας δώσουν, αλλά και να δούμε μαζί τι είναι αυτό που πρέπει να προωθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η δική μας κατεξοχήν αρμοδιότητα, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας με άλλες περιοχές του κόσμου, με διεθνείς οργανισμούς, για να αναδείξουμε το θέμα και να προωθήσουμε πολιτικές ε, που θα αποτελούν μια πρόκληση για την κοινωνία και για την οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω και εγώ τις ε, εισηγήσει σήμερα πως έχουν διαρθρωθεί, ανέφερε ήδη η Πρόεδρος, το πρόγραμμα το σημερινό και θα είναι πολύτιμες και οι εισηγήσει και τα συμπεράσματα του διαλόγου που θα επακολουθήσει για την έκθεση που έχω αναλάβει να εκπονήσω ε, εκ μέρους της, εξ της ε, Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Κράτσα για την εισήγηση αυτή και γιατί υπενθυμίσατε τους στόχους και τις ευχές της Επιτροπής μας και αυτά που ελπίζετε από την πρωτοβουλία μας. Στόχος φυσικά είναι η ενδυνάμωση της επιρροής του ρόλου των γυναικών. Προτείνω τώρα να ακούσουμε τους ομιλητές. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπουμε ένα τέταρτο το πολύ αναομιλήτρια και θα δώσω το λόγο κατά πρώτον εξ ονόματος της Επιτροπής μας βέβαια στην κυρία Βέρτ. που είναι υπεύθυνη της υπηρεσίας ίσων δικαιωμάτων και εργασίας στη Βελγική Προεδρία. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ζωέλ Μιλκέ μου ανέθεσε να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και θα ήθελε να ζητήσει συγνώμη διότι βρίσκεται, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με την πολιτική επικαιρότητα το οποίο είναι ιδιαίτερα ε, βαρύ και γι' αυτό μου ανέθεσε η Υπουργός Απασχόλησης και Ίσων Ευκαιριών να σας διαβιβάσω ορισμένα μηνύματα. Καταρχήν, ορισμένες, δια, ορισμένες ε, διαβεβαιώσεις. Ορισμένες διαπιστώσεις. Παρά το λοιπόν. γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν τα επαγγελματικά προσόντα, υπάρχουν ανισορροπίες στην εκπροσώπησή τους σε υψηλές θέσεις είτε στον πολιτικό τομέα, είτε στον, τομέα της, στον πολιτικό τομέα ή στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, στα ΜΜΕ, στα πανεπιστήμια και τις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις και στην εργοδοσία. Οι γυναίκες εκπροσωπούν το 32% των θέσεων διευθυνόντων συμβούλων, 10% των μελών των διοικητικών συμβουλίων, των περισσότερων επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο, 25% στη δημόσια διοίκηση και 4% της 100 μόνο είναι πρόεδροι μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καμία γυναίκα ε, δεν ε, είναι ε, διοικητής τράπεζας. Επίσης, οι γυναίκες δεσπόζουν στις θέσεις που δεν πληρώνονται καλά, υποπληρώνονται. Και όταν κατέχουν μία υψηλή θέση, αφορά τομείς που είναι ίσονος σημασίας από οικονομικής πλευράς, δηλαδή τον μη αγοραίο τομέα. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που προσδιαρίζουν τη διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό το διαπιστώνουμε στους τομείς όπου προεξάρχοντα ρόλο έχουν οι άνδρες. για την Βελγική Προεδρία, για την Υπουργό Απασχόλησης, αυτό το θέμα της εκπροσώπησης θα πρέπει να καταπολεμηθεί και ρυθμιστικά, από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, διότι όπως γνωρίζετε η δήλωση του Πεκίνου του 1995 προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις, ο δημόσιος φορέας, οι μη κυβερνητικές θα έπρεπε να ε, ε, δράσουν άμεσα για να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα έτσι ώστε οι γυναίκες να βρεθούν σε θέσεις αποφασιστικής σημασίας. Αυτό αφορούσε τη δήλωση του Πεκίνου το 1995. Αυτή η διαφορετική εκπροσώπηση σε θέσεις μεγάλης ευθύνης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από οικονομικής πλευράς και όχι μόνο νομικής. Διαπιστώνουμε και το βλέπουμε σε ολοένα και περισσότερες μελέτες ότι στις επιχειρήσεις που υπάρχει καλή κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών, αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα και στον χρηματοοικονομικό τομέα και στον οργανωτικό τομέα ή των δημοσίων σχέσεων. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η Υπουργός μου ε, ζήτησε να σας διαβιβάσω ορισμένα μηνύματα ως προς το ε, τρόπο δράσης. Και το πρώτο στοιχείο έγκυται στο εξής. Η άνηση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών αφορά πολλούς παράγοντες που είναι αλληλένδετοι. Υπάρχουν έμεση παράγοντες διακρίσεων καθώς και διαρθρωτικοί παράγοντες. Και αυτό αφορά το νομοθετικό, νομικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νομική πλαισίωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν θα δράσουμε λοιπόν μόνο με βάση συγκεκριμένες στοχοθετήσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα συνολικό όραμα ως προς την στρατηγική μας και προγράμματα δράσης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε οκτώ σημεία θα πρέπει να εκπονήσουμε μία στρατηγική δράση η οποία να καταπολεμήσει τα αίτια της ανισότητας και της ε, υποεκπροσώπησης των γυναικών. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο δράσης είναι να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση με δεσμευτικές δράσεις. Στο Βέλγιο συστάθηκε μία ομάδα εργασίας για να προετοιμάσει προτάσεις για ε, δημιούργηση ποσοστώσεων, εν τρίτον δηλαδή γυναίκες, στα διοικητικά συμβούλια, στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, αλλά και, στα, και ως διευθυντικά στελέχη αυτών των επιχειρήσεων. Είναι ένα επίμαχο θέμα, το οποίο ακούσαμε και χτες κατά την Υπουργική Διάσκεψη ισότητας ανδρών γυναικών που ασχολήθηκε με το θέμα της ενίσχυσης των δράσεων των κρατών μελών συζητήθηκε το θέμα των ποσοστώσεων και είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις ανάλογα με το ποια εθνική αντιπροσωπεία εκφράζεται και η συνάδελφος θα μιλήσει για το θέμα πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις και η εμπειρία τους είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, δεσμευτικά μέτρα για την εκπροσώπηση των γυναικών. Ένα τρίτο σημείο δράσης αφορά την βελτίωση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Για άλλη μια φορά τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Γιατί το ε, καθοριστικό σημείο στα διαδρομία της γυναίκας χρονικά είναι γύρω στα 30 της χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη ότι οι γυναίκες μεταξύ 30 και 40 εκείνη τη στιγμή επιλέγουν μερική απασχόληση και αυτό αφορά ένα 40% των γυναικών σε μια κοινωνία όπου ε, δίνουμε σημασία στην εργασία, η διακοπή στα σταδιοδρομίας και μέσω μερικής απασχόλησης αποτελεί ένα πραγματικό εμπόδιο έτσι ώστε η γυναίκα να κατέχει διευθύνουσες θέσεις. Για να συμφιλιώσουμε λοιπόν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή υπάρχουν ε, σημεία δράσης. Καταρχήν βρεφονιπιακή σταθμή, καθώς και άδειε μητρότητας ή πατρότητας, ενθαρρύνοντας και, τους, και τον πατέρα να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι άντρες και οι γυναίκες ε, καλύπτουν συγκεκριμένους ρόλους οι γυναίκες συμμετέχουν σε τομείς που δεν αξιολογούνται ιδιαίτερα ψηλά Αυτά τα στερεότυπα οδηγούν στην υποτίμηση των επαγγελματικών προσόντων των γυναικών. Πολλές φορές λέγεται ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να κατέχουν διευθυντικές oh. θέσεις, είναι πιο ευάλωτες, δεν μπορούν να κατέχουν τέτοιες θέσεις και αυτό ε, αποκαλύπτει τα στερεότυπα που ε, αφορούν τη σταδιοδρομία των γυναικών. Όπως σας είπα χτες, η Βελική Προεδρία διοργάνωσε μια διάσκεψη για τις μισθολογικές διαφορές και μιλήσαμε για τα αίτια αυτών των ε, διαφορών όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ένας ε, πολιτισμικός αποκλισμός και είναι δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Η Υπουργός επίσης έχει υπενθυμίσει πλιστάκης ότι η καταπολέμηση των στερεοτύπων θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην πολιτική απασχόλησης που σχετίζεται με τις νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς έχει η πράσινη ή η λευκή απασχόληση, λέει η ομιλήτρια, δηλαδή δηλαδη αυτή πολλές πολλές φορές υποεκπροσωπούνται στην πράσινη απασχόληση σε ε, εργασίες τεχνολογιών εχμής. Και αυτό αφορά και τον ε, τριτογενή τομέα. Επίσης υπάρχουν μισθολογικές ε, διαφορές και σε υψηλές θέσεις. Ως προς τις μισθολογικές διαφορές βλέπουμε ότι είναι της τάξης του 18% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένας από τους λόγους που οθεί τις γυναίκες να θυσιάζονται επαγγελματικά και να μην έχουν πρόσβαση σε ε, θέσεις ιδιαίτερα υπεύθυνε. Η Βελική Προεδρία ασχολήθηκε πραγματικά με αυτό το θέμα. Προετοιμάζουμε συμπεράσματα που θα προβάλλουμε στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του ε, Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να τονίσουμε ότι χρειάζονται στρατηγικές για να καταπολεμήσουμε αυτούς τους πολλαπλούς παράγοντες καθώς και στοχοθετημένες δράσεις. Ένα έκτο σημείο ε, Εδώ αναφέρομαι στο πρόγραμμα δράσης Επιτροπής που υποβλήθηκε στην αρχή του έτους. Υπάρχει μια πρόταση σε σχέση με τις ε, πρωτοβουλίες εποπτείας γιατί ξέρουμε ότι στον ε, επιχειρηματικό κόσμο οι γυναίκες δεν ευεργετούνται τόσο πολύ όσο οι άνδρες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των ε, γυναικών σε όλα τα δίκτυα και βλέπουμε ότι αυτή η πλαισίωση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις, για να έχουν πρόσβαση σε ε, υψηλές θέσεις και οι γυναίκες συμμετέχουν πολύ λιγότερα. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει και σε αυτό το τομέα και το 8 σημείο είναι η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρά οικονομικό φαινόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Eh, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω την σημασία ε, αυτής της ε, αιτιακής καθαρά διαφοροποίησης η οποία απορρέει και επεξήγει την κατάσταση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Άρνη Χολ από την Νορβηγία που είναι Γενική Διευθύντρια του ε, Τμήματος Σώτας Ανδρών Γυναικών στη Νορβηγία. Η κυρία Βέστριν δυστυχώς δεν είναι παρούσα και η κυρία Χολ θα λάβει το λόγο εξ ονόματός της. Θα μας πει πώς έχει η κατάσταση στη Νορβηγία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Εύα Μπρίτ και τη Ρόδη που μας κάλεσαν, ενώ δεν είμαστε κράτος μέλος, για να έρθουμε σε αυτή την ακρόαση. Επίσης, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υπουργού μου, ενός νεαρού άντρα, στην Επιτροπή σας, ο οποίος θα ήθελε να είναι εδώ πέρα, γιατί πραγματικά τον απασχολεί πάρα πολύ η ισότητα, αλλά σε λίγες μέρες θα πάρει τετρα... τετράμινη άδεια πατρότητας. Οπότε έστειλε εμένα. Τώρα, καμία χώρα δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την ισότητα ως κλειδί στην οικονομική σταθερότητα, και ανοτομία και ανάπτυξη. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Έχουμε ενδείξεις που βασίζονται στην έρευνα. Αυτά τα οποία ακούγονται στην Νορβηγία είναι το εξή. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της οικονομίας. 82% του εθνικού μας πλούτου. Το πετρέλαιο 7%. Οπότε είναι σημαντικό για εμάς το πώς χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους και πώς θα επιτύχουμε πραγματική και ουσιαστική ισότητα. Βεβαίω οι παραδόσεις πεθαίνουν γρήγορα και κάποιες φορές χρειάζεται κάποια δράση νομοθετική για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Να σας δώσω μία σύντομη εικόνα των νόμων περί ποσοστώσεων που έχουμε στην Νορβηγία τα τελευταία 25 χρόνια. Πολλά γραφεία στην ε, Νορβηγία πίστευαν ότι έπρεπε να ληφθούν νομοθετικά μέτρα και ποσοστώσεις. Οι ποσοστώσεις ξεκίνησαν από τα πολιτικά κόμματα εθελοντικά. Σήμερα έχουμε ισότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο, 40% γυναίκες στο Κοινοβούλιο και 38% στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά δεν υπάρχει νόμος περί ισότητας στις εκλογές, πρέπει να το τονίσω αυτό. Το 1988 αλλάξαμε την νομοθεσία περί και είπαμε πως 40% θα πρέπει να εκπροσωπεί το κάθε φύλλο σε όλες τις επιτροπές αντιπροσωπείες που διορίζει το κράτος. Αυτό σημαίνει πολλά και υπάρχουν και κυρώσεις. Το 1993 είχαμε αυτό το 60-40, το ίδιο δηλαδή το 40% του κάθε φύλλου για τα εκλεγμένα δημοτικά συμβούλια. Το 1993 το κάναμε δια νόμου το θέμα της γονικής άδειας, η οποία δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στην ε, μητέρα. Του χρόνου λοιπόν ε, θα γίνει 12 εβδομάδες και συνολικά η περίοδος αυτή είναι 40 εβδομάδες με 100% μισθό. Κάτι το οποίο έχει οδηγήσει βεβαίως τις επιχειρήσεις ε, σε ε, αλλαγή νοοτροπία και του γονείς. Δηλαδή το να φροντίζει κανεί τα παιδιά του είναι κάτι φυσιολογικό. Κυρώσεις υπάρχουν, λογοδοσία και η λογοδοσία είναι το βασικό. Το 2003 τέσσερις διαφορετικοί νόμοι τροποποιήθηκαν που αφορούσαν τις επιχειρήσεις για το 40% στο ΔΣ των επιχειρήσεων. Όχι για τις δουλειές, αλλά για εισηγμένε στο χρηματιστήριο εταιρείε ο, κανονισμό, ψηφίστηκε το 2006 με μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. Το Εθνικό Αρχείο Επιχειρήσεων εφαρμόζει του κανόνες ε, και οι κυρώσει φτάνουν μέχρι τη διάλυση τη εταιρεία. Το κάναμε αυτό το 2003 και ήμουν προσωπικά υπεύθυνη για τη σύνταξη αυτών των νόμων και τότε οι γυναίκες απουσίαζαν από τα διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων εταιριών. Ήταν ένα 7%. Τώρα έχουμε φτάσει στο 40,2%. Τίποτα δεν είχε γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, πριν το 2003. Η κατάσταση ήταν ντοπιαστική για όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην ενός. Είχαμε επενδύσει δισεκατομμύρια στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Η κόρες μας όμως δεν έφταναν στα διοικητικά συμβούλια, κάτι το οποίο δεν ήταν λογικό, ούτε και από οικονομική σκοπιά. Είναι θέμα απόδοσης της επένδυσης. Οι νομικές προτάσεις βεβαίως δημιουργήσαν πολλές τεταμένες συζητήσεις στα ΜΜΕ και βεβαίως εμείς από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου χρησιμοποίησαμε αυτή την κατάσταση για να προσκαλέσουμε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους για να συζητήσουν την ισότητα. Εκεί ήταν η ευκαιρία μας. Ο νόμος προτάθηκε από φιλελεύθερο συντηρητικό Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την τότε αντιπολίτευση το 2003, οπότε ήταν πραγματικά διακομματικός πλήν ενός κόμματος. Mm. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή στην ιστορία. Το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο περίμενε δύο χρόνια πριν εφαρμοστεί ο νόμος ε, γιατί περιμέναμε το βασιλιά βεβαίως, έτσι, σε μας και ήλπιζαν πως οι επιχειρήσεις θα τα κανόνιζαν μόνες τους. Οπότε έγιναν οι μετρήσεις το 2005 και τίποτα δεν είχε γίνει. Έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος και το Υπουργικό Συμβούλιο πήγε στον Βασιλιά 1η Ιανουαρίου 2006 και εφαρμόστηκε ο νόμος. Αυτό ήταν ένα μάθημα γιατί θεωρούσαμε πως με τον νόμο ως απειλή οι επιχειρήσεις θα έκαναν κάτι αλλά δεν το έκαναν. Βεβαίως στις επιχειρήσεις οι ποσοστώσεις χρησιμοποιούνται όπου είναι, έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με μεγάλη διασπορά μετοχών. Δεν ασχοληθήκαμε με τις 160.000 επιχειρήσεις σε ιδιωτικά χέρια, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως δεν υπάρχουν στις δουλειές ε, της διοίκησης ποσοστώσεις. Στον δε κρατικό τομέα οι γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση είναι 27%, μόνο 17% γυναίκες στις ανώτατες θέσεις των επιχειρήσεων συνολικά, σε όλων των ειδών της εταιρείας. Αλλά είναι αρκετά καλό το ποσοστό. Πριν από λίγα χρόνια ήμασταν στο 10%, οπότε έχει αποτελέσματα ο νόμος. Αυτό είναι σημαντικό. Κινούνται τα πράγματα. Το να είναι κανείς μέλος δοσού είναι βεβαίως μία τιμή για οποιονδήποτε άντρα ή γυναίκα και βεβαίως καθιστά τις γυναίκες πιο ορατές και επιλέξιμες και για άλλες θέσεις. Αλλά πρέπει να επενέσουμε αυτούς που πρέπει να επενεθούν. Από όταν πέρασε ο νόμος από το Κοινοβούλιο πριν εφαρμοστεί, δύο ενώσεις επιχειρηματικές έφτιαξαν προγράμματα το 2004 και το 2005 που λέγονταν θηλυκό μέλλον και φουτούρα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών για να εκπαιδεύσουν γυναίκες και άντρες για το στρατηγικό έργο που επιτελείται στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά ξεκίνησαν βεβαίω μόλις πέρασε ο νόμος από το Κοινοβούλιο και αυτό είναι σημαντικό. Και βεβαίω έχουμε πολλά τέτοια προγράμματα και στο δημόσιο τομέα, πολλά προγράμματα με μέντορες, με στόχους ε, κτλ. Αλλά δεν θα περάσω σε αυτά. Δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους ε, λάβαμε νομοθετικά μέτρα. Ε, η ποσόστοση δεν μ' αρέσει τόσο. Εν πάση περιπτώσει. Ή ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξάρτητος, φίλους, ανεξάρτητος φίλου είναι θέμα δημοκρατίας, αλλά ίσως οι ποσοστώσεις χρειάζονται για να έχουμε ίδια αποτελέσματα. Αποτελέσματα, όχι μόνο τη γιούρα ισότητα. Δεύτερον, όπως σας είπα, είναι και λογικό από οικονομική σκοπιά. Το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει ζωτική σημασία και μια ανταγωνιστική οικονομία χρειάζεται όλα τα ταλέντα ανεξαρτήτως φύλου. Έτσι, ο εξυγχρονισμός στην Ευρώπη απαιτεί την ποικιλία και μπορούμε να περάσουμε και σε άλλες μορφές ποικιλομορφίας, αλλά μένουμε εκεί προς το παρόν. Εάν συνδυαστούν λοιπόν αυτές τις πολιτικές ισότητες με τους νέους νόμους περί γονικής άδειας ε, και άδειας πατρότητας και βεβαίως πλήρη κάλυψη στην φροντίδα των παιδιών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να επιταχύνουμε τις εξελίξεις με τις ποσοστώσεις. Αλλά ίσως βεβαίως μια ποσόστοση να μην λειτουργούσε εκτός εάν οι γυναίκες ήταν ήδη ορατές αν θέλετε και διαθέσιμες και ικανές και στην αγορά εργασίας. 80% των γυναικών στην Νορβηγία εργάζονται και έχουμε παρόλα αυτά τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό γονιμότητας, ποστό γονιμότητας στην Ευρώπη, το οποίο επίσης χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε τελειώσει να πω κάποια πράγματα για τις προκλήσεις μας. Το μισθολογικό χάσμα για δουλειά ίδιας αξίας, μιλάω ανά ώρα, το ανέφερα χτες στις δύο παρεμβάσεις μου, υπάρχει. Επίσης υπάρχει διαχωρισμός και οριζόντιος και κάθετος. Υψηλός αριθμός γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Επίσης, όπως είπα, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα σχολεία, στο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να ερευνήσουμε, να επενδύσουμε περισσότερο στο να ασχοληθούν και οι άντρες και τα αγόρια στα θέματα ισότητας. Και τέλος η βία στο σπίτι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην ορβηγική κοινωνία. Χτυπά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, αλλά δεν θα επεκταθώ. Η στρατηγική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ισότητα των δύο φύλων ε, και οι συζητήσεις αυτές ορίζουν το μέλλον της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία με την ε, Κομισιόν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη και σας υπόσχομαι, σας διαβεβαιώ, πως ε, το φθινόπωρο ή μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα έχουμε έρευνες ποιοτικέ ανεξάρτητες για το τι συνέβη σε επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή του νόμου στόσεων για τη λήψη αποφάσεων. Και ευχαρίστω να τα μοιραστούμε μαζί σας. Το θέμα είναι περισσότερη ελευθερία για όλους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, για να βελτιωθεί η οικονομία και ο πλούτος της κοινωνίας και βέβαιως να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και να υπάρξει ισότητα. Όπως ξέρετε βεβαίως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση, η Ένωση τη Κοινοτομία, που στόχο έχει να δημιουργήσει 3,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2025, είναι ένα χρυσό, μια χρυσή ευκαιρία. Όπως είπε η κυρία Κουίν, η επίτροπο, εάν δεν δημιουργήσουμε καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομίε μα θα εξασθενήσουν τρομερά και θα χάσουμε ιδέε και ταλέντα. Οπότε θα πρέπει να ενσωματώσουμε την ισότητα των φύλων σε αυτή την προοπτική, καθώς επίσης και την πρωτοβουλία που έχουμε για τις πολιτικές νεότητας, την νεότητα κινήσει δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την περιγραφή αυτή των εμπειριών σας στην Νορβηγία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε μπροστά μας και τις αξιολογήσεις που κάνατε εσείς επιτόπου. Τονίζω δε ότι η συμμετοχή του, των ανδρών στα προγράμματα ισότητας των φύλων είναι κάτι το σημαντικό επίσης και το ότι ε, άνδρας είναι υπεύθυνο για το Υπουργείο Ισότητας και παίρνει τετράμινη άδεια πατρότητας δείχνει ακριβώς ότι και οι άνδρες συμμετέχουν στον αγώνα αυτών. Και τώρα καλωσορίζω την κυρία Μαριτζό Τσίμερμαν που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για την ισότητα των φύλων στη Γαλλική Βουλή. Ορίστε κυρία Τσίμερμαν έχει εργαστεί πολύ στη Γαλλική Βουλή ακριβώς για να υπάρξει κάποτε κάποια νομοθεσία υπέρ της ισότητας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα την εκπρόσωπο της Νορβηγίας την οποία είχα συναντήσει όταν είχαμε πάει στην Νορβηγία για να πάρουμε συμβουλές και να δείξουμε και εμείς τη δική μας εμπειρία στη Γαλλία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νομοσχέδιό μας, το δικό μου και του Ζαν Φρανσουά Κοπέ, είχε περάσει στη Βουλή τον Ιανουάριο, τώρα βρίσκεται στη Γερουσία και όταν εγκριθεί και από τα δύο σώματα θα γίνει νόμος. Νομίζω ότι η συνάντηση με όλους τους, τους νορβηγικούς παράγοντες τον Ιούνιο μας βοήθησε πολύ γιατί ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι είναι σωστός και δίκαιος ο νόμος αυτός Είχα την ευκαιρία στη Γαλλία και την τύχη να έχω δίπλα μου τον πρόεδρο της ομάδας μου, τον Ιωάννη Φραγκίσκο Κοπέ. Και μαζί πιέσαμε και τις επιχειρήσεις αλλά και τη Γερουσία για να εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ήταν προφανές ότι θα μπορούσαμε να το περάσουμε στη Γαλλία όπου 40% των ε, διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει, αυτό προκύπτει μάλλον από μακρά ιστορία. Υπήρξαν πολλές φάσεις και μας το είπε αυτό και η Νορβηγία ότι υπάρχουν φάσεις, δηλαδή και προσωπική ιστορία, αλλά θα ήθελα να πω ότι ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις γυναίκες Ξέρω ότι η επαγγελματική ισότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό πράγμα, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να πετύχει κανείς την ισότητα αυτήν. Είτε να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία, εδώ στη Γαλλία είναι ο έκτος νόμος περί ισότητας, είτε να υπάρχουν ποσοστώσεις και ποιώσεις ε, για μεγαλύτερη συμπερίληψη γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Η δική σας εμπειρία μας βοήθησε να επεκτείνουμε τις προτάσεις μας και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων αλλά και συνδικάτων κλπ. Στην Νορβηγία δηλαδή έμαθα ότι όταν τα πράγματα δεν κινούνται όταν αρχίζουν από τα κάτω μπορεί να αναλυφθούν πρωτοβουλίες από τα επάνω. Αυτά τα 40% δηλαδή πρέπει κάπου να τα βρούμε ακόμη και αν χρειαστούν γι' αυτό διορισμοί, θεσμικοί διορισμοί όπου μπαίνουν γυναίκες καμιά φορά σε μερικές θέσεις χωρίς να το αξίζουν απολύτως στην πρώτη φάση τουλάχιστον αλλά στη συνέχεια θα συνεχίσει η διαδικασία από τα κάτω. Και πάνω απ' όλα σήμερα τώρα που συναντώ μεγάλους επιχειρησιακούς ομίλους γαλλικούς και διεθνείς μου λένε όλοι ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μια όθηση στο σύστημα και προωθεί τις γυναίκες σε ανώτατες θέσεις. Θα σας πω τι ακριβώς λέει, το, τι περίπου μάλλον λέει το νομοσχέδιο, για να δείτε πώς προχωράνε τα πράγματα στη Γαλλία, καταρχάς υπήρξε μία θεσμική μεταρρύθμιση το 2008, δηλαδή το Σύνταγμά μας επέτρεπε την εφαρμογή ποσοστώσεων στον πολιτικό κόσμο, αλλά όχι στον επιχειρησιακό, στον οικονομικό και βιομηχανικό κόσμο. Το 2008 λοιπόν, με πρωτοβουλία της αντιπροσωπείας μας, καταφέραμε να ενδυναμώσουμε τη γαλλική νομοθεσία σχετικά και να επιτρέψει αυτή ποσοστώσεις και σε οικονομικές και κοινωνικές θέσεις. Και έτσι μπορέσαμε να νομοθετήσουμε για την παρουσία γυναικών γενικά στις θέσεις εξουσίας, διότι τα διοικητικά συμβούλια είναι ακριβώς ο χώρος όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, όπου γίνεται όλη η ανάλυση, η σκέψη, η στρατηγική καταστρώνεται μιας επιχείρησης. Και εδώ και αρκετά χρόνια σχημάτισα την πεποίθηση ότι η διαχείριση από ένα και μόνο φύλλο δεν είναι ισορροπημένη. Ενώ μία μεικτή διαχείριση επιτρέπει μεγαλύτερη ισορροπία στην διαχείριση. Το περιεχόμενο λοιπόν του νομοσχεδίου από την πλευρά των υποχρεώσεων 40% των διοικητικών θέσεων στα συμβούλια πρέπει να είναι γυναίκες, όπως στην Νορβηγία, γιατί ο πρόεδρος της ομάδας μας Ιωάννης Φραγκίσκος Κοπέ είχε ζητήσει 50% αλλά στην Νορβηγία κατάλαβα ότι πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο, ότι το 40% αφήνει περιθώριο, ενώ αν βάλουμε κατευθείαν το 50% δεν υπάρχει περιθώριο. Η ελαστικότητα λοιπόν αυτό το 40% μέσα σε έξι χρόνια από την θέση του νόμου ενισχύει. Από 1η Ιανουαρίου λοιπόν 11 θα αρχίσει να ισχύει και σε έξι χρόνια πρέπει να υπάρχουν 40% γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Στη μέση της περίοδου αυτής προβλέψαμε να επιτευχθεί το 20%. Τώρα το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου αυτού στη Βουλή είχαμε πάρει υπόψη μας τις επιχειρήσεις που μπήκαν στο χρηματιστήριο, δημόσιους οργανισμούς και ιδρύματα όπου έχει μετοχές το κράτος και έτσι διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου. Σήμερα ψηφίζουν οι γερουσιαστές αυτή τη διεύρυνση. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο γιατί δείχνει ότι όταν από τη στιγμή που αρχίσει μια διαδικασία μπορεί κανείς να προωθήσει τα πράγματα, να προχωρήσει την ιδέα πιο πέρα από ό,τι στην αρχή της διαδικασίας. Και η συνάδελφός μου που θα εισηγηθεί το απόγευμα την ψηφοφορία αυτή μας είχε πει ότι και οι εταιρείε όχι μόνο που είναι στο χρηματιστήριο αλλά που έχουν πάνω από 60 υπαλλήλου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ποσόστοση αυτή 2.000 επιχειρήσεις περίπου. 40% λοιπόν γυναικών στα διοικητικά του συμβούλια. Για τις κυρώσεις τώρα, εδώ δεν υπήρξαμε τόσο αυστηρίωσο στην Ορβηγία γιατί η μεταβατική περίοδο ακυρώνονται οι διορισμοί αν δεν πληρέεται η ποσόστοση και αυτό σε τρία και σε έξι χρόνια. Και στο τέλος και εδώ η Γερουσία προχώρησε τα πράγματα ότι θα ακυρώνονται και οι πληρωμές των κακώς διοριστέντων για να πάψουν οι διορισμοί. και ότι θα παίρνουν και παρουσίες. Από την άλλη, στην φιλοσοφία, για να το πω έτσι, του νομοσχεδίου αυτού, πρέπει να ξέρουμε ότι ο βολονταρισμός είναι κάτι σημαντικό αλλά ανεπαρκές. Γιατί αν έχει κανείς τη θέληση να δηλώσει ότι μέσα σε 6 χρόνια θα φτάσουμε το 40% καλό είναι μένα, αλλά αν δεν υπάρξει νόμος που να επιβάλλει και κυρώσεις αν δεν επιτευχθεί το 40% τότε δεν έχει νόημα το νομοσχέδιο. Παράδειγμα, το 2006 είχα περάσει ορισμένα άρθρα ενός νόμου για την επαγγελματική ισότητα όπου ζητούσα 20% γυναίκες. Τα άρθρα αυτά όμως ακυρώθηκαν από το συνταγματικό δικαστήριο και γι' αυτό έγινε η συνταγματική μεταρρύθμιση. Το ωραίο είναι ότι ο νόμος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2006. Το Δεκέμβριο 2009 περάσαμε από 9% γυναικών στα διοικητικά συμβούλια στο 8% το 2010. Αντί να προχωρούμε δηλαδή, ενώ είχαν ακυρωθεί τα άρθρα κτλ, ε, έγινε παρόλα αυτά μία πρόοδος. Σήμερα ψήφισε η Βουλή αυτό το νομοσχέδιο που σας ανέφερα και τον Ιούνιο τα διοικητικά συμβούλια έφτασαν στο 14% γυναικών ήδη χωρίς να ακόμη να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Απλό και μόνο με την σπάθα του δαμοκλέους του επικρεμαμένου νομοσχεδίου πέρασε το ποσοστό από 9 σε 14%. Αυτό δείχνει ότι πράγματι οι νόμοι πρέπει να είναι δεσμευτικοί. Εγώ χρειάστηκα πολύ χρόνο για να, μέχρι να καταλάβω ότι μόνο έτσι γίνεται πρόοδος, αλλά τώρα επίστηκα. Χωρίς νόμο δεν υπάρχει πρόοδο, δεν γίνεται πρόοδος. Και πρέπει να έχει και κυρώσεις γιατί αλλιώς ξεχνιούνται οι νόμοι. Λοιπόν, ο στόχος τώρα, πολλές φορές στη Γαλλία μια επίκριση που ακούγεται είναι ότι οι πρώτοι που θα διοριστούν μεταξύ τον Ιανουάριο, που διορίστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου δεν ήταν γυναίκες ε, που όντως ε, προέρχονταν από την επιχείρηση που είχαν τα κατάλληλα προσόντα ή κατάρτιση. Πράγματι, μερικές δεν τα είχαν, αλλά εμείς θέλουμε στα διοικητικά συμβούλια να καταλήξουμε σε ικανές γυναίκες, σε γυναίκες που να έχουν τα απαραίτητα διπλώματα και προσόντα, για να μπορούν να θεωρηθούν και τυπικά ως διοικητικοί υπάλληλοι. Και εδώ η Νορβηγία μας έδωσε την έμπνευση, χρειάζεται μία κατάρτιση Θυμάμαι όταν πήγα στην Νορβηγία ότι μας είπατε ότι προηγουμένως δεν υπήρχε σχετική κατάρτιση γιατί ένας άντρας μπορούσε να θεωρηθεί διοικητικός χωρίς ειδικά προσόντα ενώ για τη γυναίκα χρειάζεται κατάρτιση. Έτσι όμως αυτό επιτρέπει σε όλο τον κόσμο να καταρτιστεί άντρες και γυναίκες και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν γεννιέται κανείς διοικητικός ούτε διοικητικά μπορεί να επιμορφωθεί. Και έτσι δίνεται ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην αξία του διοικητικού υπαλλήλου. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι γιατί είναι απαραίτητε οι ποσοστώσεις. Λοιπόν, πάλι στην Νορβηγία είχα συναντήσει τον υπουργό σας, τον κύριο Γκαβρίλσεν, που είχε την πρωτοβουλία του νόμου αυτού και που δεν ήταν πολιτικής προελεύσεως, αλλά που είχε καταλάβει πολύ γρήγορα ότι τα διοικητικά συμβούλια δεν έπρεπε να παραμείνουν σύλλογοι ανδρών. Και σήμερα δεν ξέρω αν τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων τραπεζών ήταν μεικτά, αν δεν θα είχαν ληφθεί διαφορετικές αποφάσεις και δεν θα είχαμε καταλήξει ίσως στην κρίση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν δεν υπάρχει μεικτή διαχείριση δεν ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα της εξουσίας και σε δίκαια εκπροσώπηση της κοινωνίας. Σήμερα, πρέπει να είναι σαφές αυτό, οι, χώρες, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μισό του πληθυσμού. Στο Βέλγιο λέει 42%, στην Νορβηγία 40%, στη Γαλλία είμαστε 17%, στη Γερουσία 20% στο Κοινοβούλιο. Άρα δεν υπάρχει σωστή εκπροσώπηση της γαλλικής κοινωνίας με βάση τα ποσοστά σε έναν χώρο εξουσίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα σε χώρους εξουσίας όπως τα διοικητικά συμβούλια να υπάρξει πράγματι μία δίκαιη εκπροσώπηση και άρα και δίκαια και διαδικασία λήψης αποφάσεων γιατί δεν λέω ότι είναι καλύτερα ε, τα προσόντα μεγαλύτερα των γυναικών από των ανδρών αλλά υπάρχει μια συμπληρωματικότητα που δεν πρέπει να την αγνοούμε σε τέτοιους χώρους διότι υπάρχουν δεξιότητες αντρικές υπάρχουν γυναικείες και η συμπληρωματικότητά τους είναι αυτό που καθιστά την διαχείριση πραγματικά αντιπροσωπευτική. και άρα και πιο δεσμευτική για τη λήψη των αποφάσεων και την εκτέλεσή τους. Στη Γαλλία λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό το πρότυπο και θα θέλαμε σήμερα να αποτελέσουμε υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω απ' όλα θα ήθελα και κάτι άλλο. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δείξουμε πώς μπορούν οι πολιτικοί να προχωρήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσίμερμαν. Νομίζω ότι η εισήγησή σας ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και μας έδωσε πολλές πληροφορίες. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τις εθνικές εμπειρίες και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον προς αυτή τη θετική κατεύθυνση, κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε δύο εισηγήτριες μας. Στην κυρία Κώστα, που είναι σκιώδης εξ ονόματος των σοσιαλιστών και σοσιαλδημοκρατών εδώ στην Επιτροπή μας. Έχετε πέντε λεπτά. Κύριε Κώστα, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εξαιρετικές μας εισηγήτριες. Νομίζω ότι ήταν άκρη άκρος ενδιαφέρουσα αυτή η συνολική εικόνα κομβικών σημείων, διότι θίξατε ένα ευρύτατο θέμα, τονίζοντας ορισμένα ιδιαίτερα σημεία. Πρόκειται για τρεις πολύ σημαντικές εισηγήσει είτε ως προς τις ε, δεσμεύσεις της Υπουργού Απασχόλησης με τα οκτώ σημεία τα οποία θα πρέπει να ξαναδούμε και αυτό αφορά και τις ε, ε, δύο τελευταίες παρουσιάσεις και αυτό, αυτή την πρόταση νόμου που έχει γίνει νόμος στην Ορβηγία ε, εδώ και αρκετό καιρό και το ίδιο αφορά και τη Γαλλία και στην Ιταλία. Προσπαθούμε να προωθήσουμε μια τέτοια πλαισίωση, νομοθετική πλαισίωση, η οποία θα βοηθήσει ιδιαίτερα ως προς το θέμα των ποσοστώσεων. Θα πρέπει όμως το θέμα να το συνδέσουμε με δεσμεύσεις, κυρώσεις ή ευκαιρίες, ή κίνητρα. Στην Ιταλία χθες Έληφθη μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με από 500 γυναίκες που είναι ε, διευθύνουσες σύμβουλοι που ε, δημιούργησαν και ένα περιοδικό το Manager Impresa και μίλησαν όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και πώς μπορούν οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν αυτά τα παγκόσμια οικονομικά τρέντ, τα ηγετικά πρότυπα που υπάρχουν ως προς τους άνδρες και τις γυναίκες, το θέμα της πολυπολιτισμικότητας ως θετικό στοιχείο και τις νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προς τα που κινούμαστε, προς τα που κινείται η οικονομία και ούτω καθεξής βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη 2020 και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε στο επίκεντρο των σκέψεών μας και να μιλήσουμε για ένα καινοτόμο πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και μία γενναιόδορη θεώρηση για τις γυναίκες. Ως προς τα άμεσα ή έμεσα αίτια διάκρισης για την στρατηγική αυτή, νομίζω ότι υπάρχει και μία απάντηση η οποία σκιαγραφήθηκε ήδη. Δηλαδή να συνδέσουμε περισσότερο, περισσότερα από ένα αίτια. Έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή εποπτεία της μητρότητας αλλά και της πατρότητας, ε, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες, κατά τις πρώτες εβδομάδες. Υπάρχουν διακρίσεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Επίσης νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να μας βοηθήσει ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε πώς οι γυναίκες συμμετέχουν σε διευθύνουσες θέσεις είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Εμείς αρχίσαμε με ένα εγχείρημα στη χώρα μου το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Η ποσόστοση για να βελτιώσουμε την παρουσία της γυναίκας σε θέσεις αποφασιστικής σημασίας αφορά και την αρχική επιλογή. Εμείς βλέπουμε τις ποσοστώσεις που χρησιμοποιούν οι άνδρες για γυναίκες. Δηλαδή, αυτό έχει σημασία και ως προς το αριθμητικό στοιχείο, αλλά πώς γίνεται και η επιλογή. Θα μπορούσαμε να έχουμε οργανώσεις ή φορείς όπου θα είχαμε τράπεζες δεδομένων με τα γεωγραφικά όλων των γυναικών που έχουν αριστεύσει η καθεμία στον τομέα της, στην έρευνα, στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν γυναικεία λόμπι, αλλά κατά τον διορισμό θα έπρεπε να ασκηθεί μία πίεση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τράπεζες δεδομένων για να φτάσουμε σε αυτές τις ποσοστώσεις. Βεβαίως, με βάση τα βιογραφικά θα γίνουν επιλογές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα επαγγελματικά προσόντα, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να συμμετέχει. Επίσης υπάρχουν έμεσες διακρίσεις, όπως είπε η κυρία Τσίμερμαν, όταν μιλάμε για την κατάρτιση. Το 58% των γυναικών έχουν πτυχίο, έχει πτυχίο στη χώρα μου, αλλά στη συνέχεια έχει σημασία πώς ε, στοιχειοθετείται η επαγγελματική του σταδιοδρομία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το μισθολογικό χάσμα αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή ποιος κάνει την κατάρτιση, ποιος δίνει κίνητρα. Αυτό βρίσκεται έξω από το συμβατικό πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες κατάρτισης των γυναικών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πέρα από την ισότητα γενικά, θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένους ε, μηχανισμούς και διαδικασίες πέρα από τα στερεότυπα δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς για να αλλάξει η συμπεριφορά μας γενικότερα ως προς την αντιμετώπιση των γυναικών κατά τις ναι. ε, προσλήψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στην άλλη σκιώδη εισηγήτρια ε, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Εγώ μόλις έρχομαι από μια άλλη συνεδρίαση, οπότε έχω ξεχάσει τα χαρτιά μου και ζητώ συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Επειδή καθυστέρησα άκουσα μόνο λίγου από του ομιλητέ. την κυρία από την Νορβηγία και την κυρία από την Γαλλία, χάρηκα που άκουσα αυτές τις παρουσιάσεις, γιατί έλαβα πολλές πληροφορίες και ενθαρρύνθηκα. Το γεγονός πως συζητάμε τώρα αυτή την έκθεση είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Όμω. για κάποια κράτη-μέλη, επειδή δεν θα κατονομάσουμε κράτη-μέλη και δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη ίδια, νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως πρέπει να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Τι εννοώ. Ίσως η Επιτροπή μας θα έπρεπε να οργανώσει μια εκδήλωση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως όταν είχαμε προετοιμάσει τις συζητήσεις για την ε, οδηγία για την άδεια μητρότητας. Γιατί είχαν έρθει τότε δημοσιογράφοι από παντού και οι δημοσιογράφοι από την Εστονία, τη χώρα μου, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Κανονικά τα μία δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα και ακόμα και όταν γράφουν γι' αυτό το δείχνουν από τη σκοπιά που θέλουν. Λένε πως οι γυναίκες δεν χρειάζονται ποσόστοση και δεν καταλαβαίνουν πως οι ποσοστώσεις ε, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μία μέθοδος απλά για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να τονίσω είναι πως πρέπει να αναφέρουμε κυρώσεις στην έκθεσή μας. Εάν δεν έχουμε κυρώσεις, τότε το δικαίωμα της ισότητας υπάρχει μόνο de jure, αλλά δεν θα γίνει ποτέ de facto, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Έδωσα προσοχή, εγώ και ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και 20 χρόνια από όταν έγιναν ανεξάρτητη ξανά η Εστονία και ξέρω πως εάν δεν υπάρχουν κυρώσεις κάποια πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ πράξη. Μπορούμε να διδαχτούμε από την Νορβηγία και από την Γαλλία ακόμα και πριν περάσει η νομοθεσία από τη Γερουσία βλέπουμε πως τώρα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα κράτη-μέλη που έχουν σημειώσει καλή πρόοδο και ελπίζω η πρόοδος αυτή να διανοίξει ανοίξει τον δρόμο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη γιατί σήμερα στην Εστονία έχουμε πολιτικούς από τα δεξιά κόμματα που λένε πως έχουμε νομοθεσία τι χρειάζεται επίτροπος ίσων ε, δικαιωμάτων που έχουμε εδώ και πέντε χρόνια στην Εστονία. Τώρα βεβαίω έχει εκλεγεί νέο άτομο σε αυτή τη θέση γιατί το προηγούμενο άτομο μπορούσε μόνο να κάνει συστάσεις ε, η κυρία Κίνη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο και βεβαίως χωρίς κυρώσει δεν ακούει κανείς. Και τώρα στην Εστονία ρωτάνε, μα χρειαζόμαστε επίτροπο ίσων δικαιωμάτων ίσως να είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε. Βέβαια δεν είναι πρόβλημα ιστονικό, είναι και στα άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και σε αυτά τα οποία είναι καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν πως ε, πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να γίνουν αυτές οι συζητήσεις και ίσως τα εγγόνια μας όταν ε, θα φτάσουν σε ηλικία Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως να είναι και σε ένα Διοικητικό Συμβουλίο. Και Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα αρχίζει ο γύρος της συζήτησης για τους συναδέλφους που το επιθυμούν. Η κυρία Γκουρμάη. Δύο λεπτά η κάθε μία Ορίστε κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή μου πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλες σας συμβάλατε στις επιτυχίες που σημειώθηκαν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Ρόδη γιατί νομίζω ότι η έκθεσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και η Σίλβια βέβαια και η Σίλβια. Λοιπόν, είμαι φίλη και της Άνικεν Χούτφιλτ, θυμάμαι όταν προετοιμάζατε την νομοθεσία αυτή τα νομοσχέδια τη δεκαετία του 70 είχατε αποφασίσει ότι αν συνεργαστούν άντρες και γυναίκες δεν θα αυξανόταν μόνο η γεννητικότητα αλλά και η κοινωνική περίθαλψη γενικότερα. Και τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα. Ο Υπουργός είναι, λένε, σε πατρική άδεια. αυτό δείχνει ότι τα θέματα ισότητας των φύλων ενδιαφέρουν και τους άντρες. Επίσης πολύ ενδιαφέρον το νομοσχέδιο στη Γαλλία και είναι κρίμα που δεν μπορούσε να έρθει η Υπουργός, η η Υπουργός Ζωέλ Μιλκέτ Ξέρω όμως ότι είχε ανηλυμένη υποχρέωση για πολύ σημαντικά θέματα για την συγκεκριμένη εφαρμογή των νομοθεσίων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο πολύ συντηρητικέ κυβερνήσει η Ουγγρική και η Πολωνική, που δεν έχουν ή καμία γυναίκα υπουργό ή ελάχιστες. Ενώ η καμια γυναικα υπουργο η ελαχιστε ενω η ισπανικη και η Βελγική Προεδρία έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια για τη στρατηγική του 2020 είμαι πιο επικριτική, δεν λέει και πολλά για την ισότητα των φύλων. Ενώ η στρατηγική της Λισαβόνας έλεγε ρητά ότι ενώ προηγουμένως υπήρχαν χωριστά στατιστικά στοιχεία για τους άντρες και τις γυναίκες, τώρα είναι ανακατεμένα και έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα και γι' αυτό λυπάμαι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι η ανέχεια πλήττει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες. Όταν μιλάμε βέβαια για επιχειρησιακούς κύκλους και ηγεσία, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η προκατάληψη ότι δήθεν οι γυναίκες δεν είναι ικανές για διοικητική θέση και ευτυχώς υπάρχουν και μελέτες όπως μια γαλλική που δείχνουν ότι οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι πιο ανθεκτικές. Οι άντρες δημιούργησαν την κρίση και οι γυναίκες μπορούν να τη λύσουν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκουρμάη. Κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για, την, ε, για τις θαυμάσιες ε, παρουσιάσεις σας. Ξέρετε πως είμαι Δανέζα και η Δανέζα Υπουργό Ισότητα ήταν χθε σε μια συνάντηση και είπε «Βοηθήστε με, θέλουν να περάσουν ποσοστώσει. Εγώ προτιμώ ποιότητα από τις γυναίκες». Κουίνα που μοιάζει και η λέξη με το κότας Και είναι κατά των ποσοστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να μου δώσετε επιχειρήματα. Οπότε νομίζω πως είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις αυτές. Παρακολουθώ αυτά τα οποία κάνατε στην Νορβηγία, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω πως ε, ο υπουργό Νέος όταν εισήγαγε αυτά τα μέτρα και αναρωτιέμαι αν η Νορβηγία εμπνεύστηκε από τα μέτρα τον ε, είπα τη λεγόμενη affirmative action για ή από κάτι άλλο. Α, είπατε πως απειλήσατε ακόμα και με κλείσιμο της επιχειρήσης αν δεν ε, εκπροσωπούνταν τουλάχιστον το κάθε φύλλο με 40% στο δουσού. Και ρώτησα τις Ισπανίδες ε, συναδέλφους ε, όταν πέρασαν την νομοθεσία και εκεί αν σκέφτονταν κάτι τέτοιο και είπαν όχι, γιατί έχουμε 20% ανεργία και δεν μπορούμε να πούμε πως θα κλείσουμε επιχειρήσεις, αλλά ξέρω πως η κατάσταση στην Νορβηγία είναι διαφορετική. Και τώρα στο κόμμα μου στη Δανία έχουμε την συζήτηση το ποια μέτρα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη. Στη Γαλλία ποια είναι τα μέτρα σας γιατί τη διάβαζα την νομοθεσία έξι μήνες πριν στη Μόντ, στη, στη Λιμπερασιόν, όταν ταξίδευα πήγαινε ερχόμενη από τη Σουηδία, αλλά μετά νομίζω πως η συζήτηση εξαφανίστηκε. Δυστυχώς μου λέτε πως θα ψηφίσετε την νομοθεσία αυτή στην ε, Γερουσία και ακόμα την επεξεργάζεστε. Πότε μπορούμε να περιμένουμε να περάσει αυτή η νομοθεσία. Και τέλος, για την κατάσταση στο Βέλγιο, είπατε για τα έξι μέτρα. Ε, πότε περάσατε εσείς το 30% γυναικών. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τόμψον. Η κυρία Κράτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε ήθελα να ευχαριστήσω τις συζητήτρες γιατί ήδη ήταν πολύ συγκεκριμένες και πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις τους και πολύ χρήσιμες κατά συνέπεια. Θέλω να ρωτήσω την εκπρόσωπο της ε, Υπουργού για το θέμα της ε, ε, Βελγικής Προεδρίας. Ε, μπορείτε να μας πείτε, πέρα από την εμπειρία τη Βελγική, ως Προεδρία, αν στοχεύετε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία συγκεκριμένη, αν είσαστε ήδη σε συζήτηση στο Συμβούλιο, αν τη συζητείτε με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κράτσα. Σας ε, προτείνω εδώ να φτάσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Δίνω το λόγο στην κυρία Χόλη, η οποία θα πρέπει να αποχωρήσει σε λίγο. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Χόλ. Okay. Ορίστε με μικρόφωνο. Πρέπει να φύγω για το Όσλο σε λίγο. Αλλά σας ευχαριστώ για τα εξαίρετα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Η Ιταλική πρόταση για τις τράπεζες δεδομένων με βιογραφικά. Αυτό έχει 20 χρόνια που το δοκιμάσαμε και δεν βοήθησε. Δεν βοήθησε. Δεν τα χρησιμοποίησε κανείς αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν όμως ακόμα. Ως προς τα ΣΥΠΑ, εκείνοι δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο θετικό για τον επιχειρησιακό τομέα. Εμείς εμπνευστήκαμε με τον, από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι ποσοστώσεις σε άλλους τομείς από το 1998 και μετά για δημόσιες επιτροπές και τέτοια και τα ίδια ή ανάλογα προσπαθήσαμε να κάνουμε και για τις επιχειρήσεις και τις ποσοστώσεις καθώς και για τις κρατικές επιχειρήσεις βέβαια. Και πέρυσι Εφαρμόσαμε τα ίδια και για πιο μικρές επιχειρήσεις και δήμους και κοινότητες. Όσο για τον Υπουργό μας, τι να σας πω. Εμείς ψάχνουμε τις δεξιότητες, τους καταλληλότερους, αλλά οι επιτροπές διορισμών στις μεγάλες τουλάχιστον εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν να χρησιμοποιούν και λαμπτήρες φθορισμού, όχι μόνο φακούς, λοιπόν προβολής να χρησιμοποιούν. Αυτό είναι η διαφορά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία. Λέει ο νόμος ανθρώπους με υψηλά προσόντα από ολόκληρο τον πληθυσμό, όχι μόνο το μισό. Και κάτι ακόμα, οι κυρώσεις δεν επιβάλαμε νέες κυρώσεις για την εφαρμογή του νομοσχεδίου στην Νορβηγία γιατί επί 30 χρόνια υπήρξαν κυρώσεις ώστε να γίνει σεβαστός ο νόμος για τη σύσταση των διοικητικών συμβουλίων σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Εδώ και 30 χρόνια απλώς προσθέσαμε ένα νέο κριτήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χόλ πρέπει να επιστρέψει στο Όσλο όπως, Όσλο όπως μας είπε. Τη χαιρετούμε δεόντως. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέρτς για να μας κάνει τα σχόλια και τις απαντήσεις της. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Καταρχήν, για το Βέλγιο καθεαυτόν το Design Βέλγιο. Νομίζω ότι η ανάλυση της Υπουργού ε, ήταν προσωπική και εγώ απλώς σας τη διάβασα τώρα για το τι σκοπεύει να κάνει ως υπουργό, ως Βελγίδα τα λέω αυτά, σκέφτεται το θέμα των ποσοστώσεων, την πιθανότητα των ποσοστώσεων ή άλλων θετικών και βολονταριστικών δράσεων και γι' αυτό αποφάσισε να εγκαθιδρυθούν μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στην κυβέρνηση μια ομάδα εργασίας από τις υπηρεσίες πολλών Υπουργείων που να επεξεργαστούν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Με τα παραδείγματα βέβαια και τα προηγούμενα της Νορβηγίας και της Γαλλίας το ετοιμάζει αυτό λοιπόν η κυβέρνηση. Αυτό για το Βέλγιο. Τώρα για το θέμα της Βελγικής Προεδρίας. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι η προτεραιότητα που έθεσε το Βέλγιο ως Προεδρία είναι η ισότητα των μισθών. Εδώ ετοιμάζουμε συμπεράσματα για το θέμα αυτό της μισθολογικής ισότητας που έχουν κάποια σχέση και με το θέμα μας το σημερινό στα συμπεράσματα αυτά λοιπόν προτείνουμε στα κράτη-μέλη, δεν ξέρουμε αν θα περάσει βέβαια, αλλά από αυτό που προτείνουμε είναι τα κράτη-μέλη να καθορίσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική και να αναφέρονται, να απαριθμούνται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν ρητά. Μεταξύ των μέτρων αυτών να υπάρχουν και ποσοτικά για την πρόσβαση των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις. Αυτό το προσχέδιο βέβαια κειμένου δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα αλλά πολιτικού και θα δούμε πού θα καταλήξει. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αν όλα πάνε καλά θα εγκριθεί από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ της 6ης Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου. Και θα δούμε αν θα σημειωθεί καμία πρόοδος. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία με την Βελγική Προεδρία. Έχουμε πολλά ε, ερωτήματα, πολλά κοινά ζητήματα και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εξίσου καλά και στο μέλλον. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζίμερμαν. Έχετε το λόγο. Θα σας απαντήσω εντάχει για να ισχύσει ένας νόμος θα πρέπει να περάσει από, το, ε, από την Εθνοσυνέλευση και μετά από τη Γερουσία. Σήμερα περνάει από τη Γερουσία. Θα πρέπει να μας δώσετε το χρόνο λοιπόν να τεθεί σε εφαρμογή. Θα τεθεί σε ισχύ λοιπόν από την 1η Πρώτου 2011 και μετά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, διότι μεταξύ Εθνοσυνέλευσης και Γερουσίας ε, υπήρξαν πιέσεις από την εργοδοσία για να μην ε, υπάρξει νόμος. Σήμερα θα ψηφιστεί κανονικά στη Γερουσία χωρίς μεγάλες δυσκολίες και σε δύο χρόνια μέσα σε τρία χρόνια θα δούμε κατά πόσο βρισκόμαστε στο 20%, αν όχι θα ισχύσουν οι πρώτες κυρώσεις. Σε έξι χρόνια, αν δεν είμαστε 40%, θα επιβάλλουμε τις κυρώσεις επίσης. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε 6-7 χρόνια θα φτάσουμε σε ένα 40% εκπροσώπηση γυναικών σε 2.000 επιχειρήσεις της Γαλλίας, στα διοικητικά συμβούλια, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και ε, νομίζω ότι η Βελική Προεδρία έχει, και κοινοβουλευτικές, έχει αναλάβει και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτό το πλαίσιο στα μέσα Νοεμβρίου και είναι ένα από τα θέματα που θα θίξουμε. Φαντάζομαι ότι η υπουργό σας θα το προωθήσει το θέμα, διότι όταν καλούμε το σύνολο των Ευρωπαίων συναδέλφων, τότε προσκαλούμε και τον ελόγο, την ελόγο υπουργό. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Έκανα. Ποιος είναι ο νόμος του νομοθετήματος έτσι ώστε να το βρω. είναι ο, ο, το νομοθέτημα νόμος Κοπέ Τζίμερμαν. Γιατί έβαλα πρώτο το Κοπέ. Γιατί γνωρίζετε όταν ο, η πρόεδρος της ομάδας, ο πρόεδρος ομάδας σας υποστηρίζει σε μία πρόταση νόμου, όπου γίνεται λόγος για 40% εκπροσώπηση γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος. Γι' αυτό ο νόμος φέρει το όνομα Κοπέ Τζίμερμαν. Ευχαριστούμε κυρία Τζίμερμαν και να σας ε, συγχαρώ για αυτό το μελλοντικό νόμο ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και μας ε, παρουσιάσατε την ε, γαλλική πραγματικότητα. Θα θέλαμε τώρα οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης να έρθουν εδώ δίπλα στο Προεδρείο, στην πλευρά του Προεδρείου. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ. Προτείνω να μιλήσουμε για τα απαιτούμενα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χαίρομαι που βρίσκονται εδώ τα μέλη του ΠΑΛΕΝ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τάιμα Σάμαν για να μας κάνει την ε, παρουσίασή της. Είναι διευθύντρια, όπως γνωρίζετε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Γυναικών σε ηγετικέ θέσεις. Έχετε το λόγο. Λυπάμαι γιατί ανέκυψε ένα τεχνικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Είμαι εδώ εξ του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Γυναικών σε ηγετικές θέσεις που εκπροσωπεί 100 περίπου γυναίκες, μερικές εκ των οποίων βρίσκονται στην αίθουσα που προέρχονται, που είναι Ευρωπαίες καταρχήν, προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέρχονται από τέσσερις διαφορετικούς τομείς, ε, δηλαδή από το δημόσιο τομέα, από επιχειρήσεις σε διευθυντικές θέσεις, από πανεπιστήμια και από ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική, ένα σημαντικό κενό. Είναι ε, δύσκολο για τους άνδρες να ε, βγουν από το γραφείο τους για να συναντήσουν, να πάνε να βρεθούν με τα παιδιά τους, με τον κοινωνικό τους περίγειο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις γυναίκες να τρέχουν, να φεύγουν από τα γραφεία τους για να πρέπει να ανταποκριθούν σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το δίκτυο εδώ και τρία χρόνια. Έχουμε 100 μέλη στις ΙΠΑ και σε άλλα ε, μέρη του κόσμου. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις γυναίκες, μιλάμε για τις γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις αυτό δεν σημαίνει ε, ότι βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων πάντα. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε πόσο προχωράμε ε, στη, στις κλίμακες ηγετικών θέσεων. Κάνουμε μία πρώτη διαπίστωση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Προσπαθήσαμε να βρούμε δεδομένα. Δεν υπάρχουν επαρκείς ε, μελέτες και πολλά, ε, πολύ λίγα αριθμητικά στοιχεία και όταν φτάσουμε σε επίπεδο middle management δεν υπάρχουν καθόλου αριθμητικά στοιχεία. Θα ήθελα να σας ε, διαβάσω τα διάφορα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε. Υπάρχει η βάση δεδομένων της Επιτροπής για το decision making Επίσης, στα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχουμε στοιχεία για τις γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια, αλλά όχι ως προς το middle management. Υπάρχει και η Society 21st που μας έδωσε στοιχεία. Θα πρέπει όμως να ε, καταγράψουμε ότι ε, εκλείπουν στοιχεία, λείπουν στοιχεία σε σχέση με τη θέση των γυναικών για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Μας είπατε να δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι κρατικές πολιτικές, υπάρχουν ε, ευρωπαϊκές οδηγίες που θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις χώρες για την μισθολογική ισότητα για την παιδική ηλικία και στην Ορβηγία και Γαλλία σύντομα θα έχουμε στοιχεία για τις γυναίκες στα διευθυντικά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό που έχει σημασία όμως η εφαρμογή του νόμου και η προσαρμογή του ανάλογα με την αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή ε, υπάρχουν ε, διαφορετικές θεωρήσεις του ζητήματος ως προς την έλλειψη δεδομένων αρχίσαμε, ξεκινήσαμε μία έρευνα για να δούμε πού βρίσκονται οι γυναίκες στην ιεραρχία σήμερα και να προτείνουμε κάτι το συγκεκριμένο. Υπάρχουν στοιχεία, αλλά είναι ελλειπή. Και αυτό έχει σημασία είναι να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα για να δούμε σε ποιο επίπεδο πρέπει να δράσουμε. Γίνεται μία διαπίστωση, είπαμε πολλά και δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά οι γυναίκες αποτελούν το 60% ε, των διπλωματούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μόνο 13 γυναίκες είναι επικεφαλής μεγάλων ε, οικονομικών ομίλων. Άρα το ζήτημα είναι κατά πόσο όχι μόνο κατά πόσο βρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια, αλλά κατά πόσο συμμετέχουν σε ηγετικές θέσεις. Υπάρχουν ε, μελέτες που καλύπτουν μόνο έξι κράτη-μέλη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πού βρίσκονται οι γυναίκες και πού έχουμε χάσει στοιχεία σε αυτό το μονοπάτι. Η άδεια μητρότητας δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Ξέρω ότι μόλις ε, ψηφίσατε μια πρόταση παράτασης της άδεια μητρότητας. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί φεύγουν μετά, δηλαδή επανέρχονται στη θέση εργασίας και μετά αποχωρούν. Στη μελέτη που διενεργήσαμε είδαμε ότι φεύγουν και δεν έχουν ε, αρκετή εργασία, διότι τα διευθυντικά στελέχη αλλάζουν οπτική γωνία, δηλαδή δεν έχουν πια αρκετές ευθύνες, διότι θεωρείται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευθύνες. Και θεωρώ ότι αυτό ισχύει και στον πολιτικό τομέα. Δηλαδή, αλλάζει η θεώρηση ως προς τη δυνατότητα ευθύνης. Δηλαδή θεωρούμε ότι μια γυναίκα που έχει ένα ε, βρέφος ή ένα πολύ μικρό παιδί δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στις ευθύνες της. Γι' αυτό και δεν της ανατίθεται σημαντικό έργο και αρμοδιότητες. Γιατί αποχωρούν λοιπόν και πώς μπορούμε να προωθήσουμε το ζήτημα ώστε να παραμείνουν Βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα εμπειρικά στο δίκτυο γιατί μας μίλησαν γυναίκες οι οποίες κατήχαν ηγετική θέση αρχικά αλλά στη συνέχεια δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται καταρχήν στην Νορβηγία υπάρχει μια σφαιρική θεώρηση του ζήτηματος. Μιλάμε, μιλάμε για γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια, που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία 20 με 30 χρόνια είχαμε να κάνουμε με μία συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες επανέρχονται μετά από άδεια μητρότητας, δηλαδή βλέπουμε ότι φτάνουμε σε χάσματα, δηλαδή ε, βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν εξομοιώνονται με τους άντρες, ιδιαίτερα όταν γεννήσουν. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου η ευφυΐα των γυναικών είναι πολύ γνωστή. Δηλαδή είχαμε καταρχήν τον θεσμό των παλακίδων, των κουρτιζάν, που εξελίχθηκε ανά το χρόνο μετά το 18ο αιώνα. Και βλέπουμε ότι τα πράγματα περιπλέκονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης έχουμε να κάνουμε με την επιλογή μεταξύ μητρότητας και σταδιοδρομίας. Δεν ισχύει αυτό για όλους, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Υπάρχουν στοιχεία και παραδείγματα που το επιρρονίουν αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να αναφερθούμε και στις ΗΠΑ, επικρίνουμε τη Γερμανία ιδιαίτερα, αλλά δεν τα, καταφέρει, δεν καταφέρνει και τόσο άσχημα η Γερμανία. Επίσης, έχουμε γυναίκες σε ηγετική θέση, που οι γυναίκες είναι και πολύτεκνες. Αυτό το βλέπουμε σε χώρες όπως η Νορβηγία. Στη ε, Γαλλία βλέπουμε ότι ένα 65 με 80% γυναικών με δύο παιδιά που εργάζονται. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες που απαρνούνται τη μητρότητα για να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη σταδιοδρομία. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί επιβάλλουμε μία επιλογή στις γυναίκες που δεν επιβάλλεται στους άνδρες. Δηλαδή τους λέμε πολλές φορές υπάρχει το δίλημα ή οικογένεια ή μητρότητα ή επαγγελματική σταδιοδρομία. Βλέπουμε ότι οι νόμοι για την ισότητα ή για τις θετικές διακρίσεις μπορούν να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Θα ήθελα να επανέλθω σε μια ευρωπαϊκή οδηγία που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή τη μισθολογική ισότητα, η οποία δεν έχει επιτύχει τους στόχους της, θα πρέπει να μας απασχολήσει ή τις ποσοστώσεις στα πλαίσια της ιεραρχίας. Εγώ βρίσκομαι σε μια διληματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, δεν απλουστεύεται εύκολα και θα πρέπει να δούμε πού και πώς μπορούν να βρεθούν λύσεις. Εκεί όπου δεν υπάρχουν νόμοι θετικής διάκρισης και μισθολογικής ισότητας, αν δεν υπάρχει μία πολιτική εποπτείας, τότε δεν, μπορεί να δεν μπορούν να ισχύσουν αυτά τα μέτρα, διότι μιλάμε πολύ θεωρητικά. Δεν έχουμε ε, αριθμητικά στοιχεία και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε αν δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν και δύο άλλα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το θέμα της εκπαίδευσης, μιλήσαμε για στερεότυπα που προωθούν και άνδρες και γυναίκες. Οι, τα κορίτσια και, και οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν διαφορετική, πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό διαφορετικά. δεν θα πρέπει να δεσμεύονται από αυτά τα στερεότυπα. Και υπάρχουν mm. και θετικές πολιτικές έτσι ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν στη, στα υψηλότερα κλιμάκια της εκπαίδευσης. Γιατί μόνο έτσι και τα κορίτσια μπορούν να ταυτιστούν με αυτά τα πρότυπα, έτσι ώστε να δουν ποια οδό θα ακολουθήσουν, ποια πορεία θα ακολουθήσουν. Θα πρέπει να μιλήσουμε για συνέργεια δημόσιου ιδιωτικού τομέα, διότι Θα ήθελα να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ε, έχω έργαστη και για, για μεγάλες, σε μεγάλες κοινοπραξίες ή αμερικανικές εταιρείες και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πολιτισμικό χάσμα με την Ευρώπη. Σημασία έχει ποια είναι η, ε, τι αντιπαλότητα υπάρχει και πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε αυτές τις ε, δυνάμεις. Πολλές γυναίκες στην ναι. Αμερική δύσκολα μπήκαν σε αυτά τα, τα γυναικεία δίκτυα. Αλλά δεν θα πρέπει να δεχτούμε τον πατερναλισμό που προωθείται στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει μία ε, σχέση δυνάμεων η οποία να είναι θετική. Και οι νόμοι στην Αμερική κατά των διακρίσεων βοηθούν, τις, ε, βοηθούν την προώθηση της θέσης των γυναικών ως προς τις ε, διευθυντικές θέσεις είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν γυναίκες. Διαφορετικά θα αχθούν ενώπιον δικαστήριων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική και πολιτική πίεση έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να είναι υποχρεωμένες να λάβουν θέση. Εγώ εργαζόμουν σε μία επιχείρηση μέχρι πρόσφατα στη Microsoft όπου δεν υπήρχε, ποτέ δεν υπήρχε κάποια απειλή απέναντι στις γυναίκες, αλλά αυτό που είχε σημασία είναι να, ήταν να βρεθεί ένα πλαίσιο δημιουργικότητας όπου να μπορούν να συμμετέχουν και οι γυναίκες. Δεύτερο πράγμα που δεν κάνουν αρκετά οι γυναίκες είναι η δικτυοποίηση, η δικτύωση. Δίκτυα για να ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Και υπάρχει εδώ το παράδειγμα δύο επιχειρήσεων που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυό μας ως πεδίο εσωτερικής πολιτικής για να αντιμετωπίσουν τα διευθυντικά του στελέχη έναν διαφορετικό κόσμο για να μπορέσουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες ή όπως λέμε στα φραγκοαγγλικά skills για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επιχείρηση καλύτερα. Και η πολιτική αυτή των ανθρωπίνων πόρων και στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα θέμα κλειδί. Τέλος, η εκπροσώπηση των γυναικών, μιλήσαμε για πρότυπα και ρόλους υπάρχει και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαμάν. Τώρα χαιρετίζω την παρουσία της κυρίας Ειρήνης Νατιβιδάδ, Προέδρου του Global Summit of Women. Καλώς ορίσατε. Στη συνεδρίασή μας έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Επιτροπή για ένα θέμα το οποίο μου είναι τόσο προσφυλές. Για όσες από σας δεν το ξέρετε, η Παγκόσμια Σύνοδος Γυναικών συγκεντρώνει γυναίκες από τις επιχειρήσεις και το κράτος για να δούμε πώς θα επιταχύνουμε τις ευκαιρίες των γυναικών παγκοσμίω. Υπάρχει και ένα κομμάτι μας που λέγεται «Γυναίκες Διευθύντριες» και εδώ και 20 χρόνια κάνουμε έρευνες για τις γυναίκες διευθύντριες παγκοσμίω για να δημιουργήσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες έτσι ώστε όταν λέμε δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκες να έχουμε τα ακριβή νούμερα. Όταν ξεκινήσαμε το 1998 μόνο Μία οργάνωση στον κόσμο έκανε έρευνα, Catalyst λεγότανε, στι ΗΠΑ που εξέτασε τις 500 μεγαλύτερε εταιρείε. Πρόσφατα ξεκινήσαμε μία έρευνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για να συνδυάσουμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια ανά τον κόσμο, γιατί κανείς δεν τα είχε συνδυάσει ποτέ για να έχουμε μια παγκόσμια εικόνα του που βρίσκονται οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίω. Και με έκπληξη διαπιστώσαμε πως Έχουμε πλέον δεδομένα για 51 χώρες από 26 διαφορετικές πηγές. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πω απόψε είναι κάποια από τα ευρήματα κλειδιά αυτές της έρευνας. Όχι μόνο για το πού βρίσκονται οι γυναίκες αλλά και για το τι κάνουν οι χώρες για να επιταχύνουν την παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πώς είναι η κατάσταση λοιπόν στην Ευρώπη. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες, είναι λίγο δύσκολο με τα φώτα αλλά εάν μπορείτε να τα δείτε θα δείτε πως η Ευρώπη κυμαίνεται από το 40,3% στην Νορβηγία που είναι το ανώτατο και η Σουηδία 21% μέχρι το χαμηλό το ποσοστό που είναι στην Ιταλία Πορτογαλία και Κύπρο όπου η εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια είναι γύρω στο 3% οπότε ενώ η ευρωπαϊκή ιστορία έτσι μοιάζει κάπως καλή, αν το δούμε συνολικά δεν είναι τόσο καλή η περίπτωση. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα ΣΥΓΜΑ είναι κάτω από το 20%. Όχι και πολύ σπουδαία. Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά. Εάν δείτε εκεί πέρα, η υψηλότερη στήλη είναι η Ευρώπη, με 11,9 κατά μέσο όρο. Δεν ακούγεται φοβερό, αλλά αν συνειδητοποιήσετε, συγγνώμη, συγγνώμη δεν το διακρίνω, Αυτό, α, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, κρατήστε, σβήστε τα φώτα. θα είμαστε έτσι στο σκοτάδι. Κείμενται λοιπόν από 11,9% αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως έχουμε το 40% της Νορβηγίας μέχρι το 3% στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Αν το συγκρίνουμε με την Βόρεια και Νότια Αμερική βλέπετε πως είναι 9,9%. Δηλαδή Σκεφτείτε, από το 15% στη ΣΥΠΑ που θεωρείται το υψηλότερο μέχρι το 5% στο Μεξικό. Κοιτάξτε τώρα, Ασία ειρηνικό. 6,5% μόνο από το ανώτατο 10% στις Φιλιππίνες, στη χώρα στην οποία γεννήθηκα, μέχρι το 1,4% στην Ιαπωνία. Και τελευταία περιοχή, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Από το 14% του Ισραήλ μέχρι 0,2% Σαουδική Αραβία. Εν ολίγης, δεν έχει σημασία ποιο κομμάτι του πλανήτη εξετάζουμε, αν είναι η Ευρώπη, η Αμερική, η Ιαπωνία. Η εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, ηγετικές θέσεις των επιχειρήσεων είναι ελάχιστη. Οπότε δεν είναι φοβερά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάποιος ήρωας. Ίσως Νορβηγία και Σουηδία. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί ήρωες εδώ πέρα συνολικά. Οπότε τι κάνουν οι χώρες. Ακούσατε ήδη από το προηγούμενο πάνελ τι γίνεται στην Νορβηγία και τη Γαλλία και το πώς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πιο δημοφιλή στρατηγική που είναι οι ποσοστώσεις. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Αριστερά έχουμε τις χώρες με ποσοστώσεις, οι προτινόμενες ποσοστώσεις για να καλύψουν όλες τις εταιρείες. Δηλαδή εταιρείες εισηγμένες, ε, ΑΕ μάλλον, με συγχωρείτε. Η Ισπανία επίσης, η Νορβηγία, η Ισλανδία μόλις πέρασε ένας νόμος για τις εταιρείες εισηγμένες και η Γαλλία και η Ολλανδία ε, τώρα περνάνε την νομοθεσία. Η Ολλανδία έχει κάπως δύσκολο δρόμο μπροστά της γιατί θα πρέπει να περάσει και ένα 30% στην ε, ανώτατη διοίκηση. Εάν δείτε την μέση στήλη είναι οι χώρες που έχουν ποσοστώσεις για δημόσιες και κρατικές εταιρείε. Το Ισραήλ το ξεκίνησε το 1993. Στον εταιρικό κώδικα πέρασε ένα σχετικό νόμο, Νότια Αφρική το 1996, ε, μετά το Apartheid για να μπορέσουν περισσότεροι Νότια Αφρικανοί να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα. Αλλά κοιτάξτε τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιρλανδία και την Ισλανδία ε, λυπούμε για το άτομο το οποίο γνώρισε για τη Δανία, έπρεπε να γνωρίζει πως υπάρχει ήδη ποσόστοση για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Υφίσταται ήδη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι τεράστιες. Μιλάμε για σιδηρόδρομους, ε, αεροπορικές εταιρείες, ε, εταιρείε ενέργειας, πετρελαϊκές καμιά φορά. Τώρα η Γερμανία δεν έχει στο ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά το κρατήδιο του Βερολίνου, 50% ε, Ρεμβέργη επίσης, για τις ε, εταιρείε τις δημοτικές αυτών των επιχειρήσεων ή όπου έχει μετοχές ο Δήμος. Στον Καναδά, ούτε εκεί έχουμε ομοσπονδιακή ε, νομοθεσία, αλλά η επαρχία που συνεχώς προσπαθεί να αποσχιστεί, το Κεμπέκ, έχει 50% ποσόστοση και είναι στο 40,9% ήδη. Το Βέλγιο, ακούσατε, ε, έχει κάτι που προτείνεται στο ομοσπονδιακό επίπεδο και πάλι ο Καναδάς ως πρόταση. Αυτό ήθελα να σας το δείξω για να σας δώσω μια εικόνα του ότι έχουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά βεβαίως κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν αυτό το τσουνάμι ποσοστώσεων στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα γιατί λειτουργεί. Είτε μας αρέσει η λέξη ποσόστοση είτε όχι. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε τους αριθμούς γρήγορα τότε η, η νομοθεσία λειτουργεί. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι το έκανε η Νορβηγία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίε ότι μπορεί να επιτευχθεί. Έλεγαν πως δεν βρίσκουμε γυναίκες, το έκαναν μέσα σε δύο χρόνια. Βρήκαν τις γυναίκες, όταν έλεγαν πως δεν θα βρεθούν αρκετέ γυναίκε, και έγινε χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ε, ενώ οι εταιρείε έλεγαν πως θα δημιουργηθεί χάος αν τα αναλλάξουν όλα τα δοσού αμέσω και να γίνουν 40% γυναίκες. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Τρίτον, γιατί αρέσει αυτό στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν ήδη ποσοστώσεις ως μέτρο. Οπότε περνάνε οι ποσοστώσεις από το δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Και τέλος, η Ευρώπη έχει πολλές δημόσιες εταιρείε. Δηλαδή το κράτος είναι μεγάλος μέτοχος γιατί ε, έχει πολλές μετοχές σε αυτές τις εταιρείε, οπότε ορίζει τα δουσού και την εταιρική διακυβέρνηση. Γι' αυτό σαρώνουν τώρα οι ποσοστώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειλικρινά θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορέσει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θεωρώ πως η Ευρώπη θα ξεπεράσει όχι μόνο τη ΣΥΠΑ αλλά οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο με το να αλλάξει το πρόσωπο των μελών του Δουσού και θα παίξει έναν ηγετικό ρόλο και στο πώς άλλες χώρες και οι δικοί μου θα δουν πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα ΔΣ. Μία άλλη στρατηγική και αυτή τη φορά από τον ιδιωτικό τομέα, όπως βλέπετε, έχουμε χρηματιστήρια και επιτροπές εταιρικής διακυβέρνησης που τώρα θεωρούν πως η ποικιλομορφία του ΔΣ είναι προϋπόθεση εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή απαραίτητο τμήμα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Η Φιλανδία ήταν η πρώτη χώρα το 2003 που είπε πως η ποικιλομορφία στο ΔΣ θα πρέπει να είναι στον κώδικα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Το οκτώ το ενίσχυσαν και είπαν η ποικιλομορφία του φίλου Βλέπετε εδώ πέρα το δείγμα. Φιλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη έχουν δηλώσεις στις, ε, στους εταιρικούς, εταιρικής διακυβέρνησης για αυτό το σκοπό. Τώρα οι ποσοστώσεις διαφέρουν ως προς την αυστηρότητά τους. Δηλαδή κάποιες έχουν μια υποχρέωση συμμόρφωσης που σημαίνει πως κατ' ουσίαν ντροπιάζουμε τις εταιρείε οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές γιατί ζητάμε να εξηγήσουμε γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Η Γερμανία το έχει αυτό και μόλις τώρα εγκρίθηκε αυτή η σύσταση από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και ζητάνε από τις εταιρείε να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες στην ετήσια τακτική γενική του συνέλευση. Η ΕΠΑ δεν είναι πρωτοπόρο σε αυτό. Η Επιτροπή της Κεφαλαίου Αγοράς απαιτεί τώρα να αναφέρεται στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρεία ε, η πρόοδο σε αυτό. Η πιο επιθετική πρωτοβουλία δεν είναι ευρωπαϊκή, είναι στην Αυστραλία. Αρχές του 2011 οι εταιρείε εισηγμένες στο Αυστραλιανό χρηματιστήριο πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό γυναικών στο ΔΣ, το ποσοστό γυναικών στη διοίκηση και συνολικά στο εργατικό δυναμικό και να εξηγήσουν τι σκοπεύουν να κάνουν για να αυξηθούν αυτά τα νούμερα. Αυτό είναι ίσως η πιο επιθετική πρωτοβουλία που υπάρχει σήμερα. Η τρίτη στρατηγική που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ε, αυτή την οποία θεωρώ την πιο αποτελεσματική, αναφέρθηκε πιο πριν. Αυτό το οποίο λέγεται το επιχειρηματικό επιχείρημα για τις γυναίκες στο ΔΣ. Τι λέμε κατ' όλες αυτές οι μελέτες που βλέπετε, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και όπως βλέπετε από την Τουρκία και το Βιετνάμ, καταλήγουν στο εξή αποτέλεσμα. Όσο περισσότερες γυναίκες υπάρχουν στην ανώτερη διοίκηση και στα ΔΣ εταιριών, τόσο, το καλύτερα αποτελε... τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα των εταιριών όσον αφορά την απόδοση ενεργητικού, την απόδοση επενδύσεων, την αύξηση του μερίσματος προς τους ε, μετόχους ε, και όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και τη γενικότερη εποπτεία της επιχείρησης. Οπότε υπάρχει ήδη εκτεταμένη έρευνα, ελπίζω να ήταν εδώ οι φίλοι μας από την Δανία για να ακούσει τα επιχειρήματα για τον Υπουργό της. Έχει αποδειχτεί ήδη. Το πρόβλημα είναι πως δεν ε, έχει ακουστεί πολύ στον ιδιωτικό τομέα. Πολλά πανεπιστήμια κάνουν μελέτες και ξέρετε τι κάνουν οι καθηγητές κάνουν έρευνα και λένε τι φοβερό, δημοσίευσα, έκανα άλλη μία δημοσίευσα, αλλά κανείς δεν το ξέρει. Ακούσατε τις μελέτες της McKinsey και του Catalyst, αλλά επίσης αυτοί απευθύνθηκαν και στα ΜΜΕ για να μιλήσουν για αυτό το θέμα και πράγματι τα ΜΜΕ πρέπει να ενημερώσουν τις εταιρείες ότι είναι προς το οικονομικό του συμφέρον να έχουν περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ. Δεν είναι θέμα ισότητας δικαιοσύνης ούτε καν επένδυσης στην εκπαίδευση, αλλά θέμα απόδοσης της επένδυσης στην ίδια του στην εταιρεία. Να τελειώσω λέγοντας το εξής. Τι θα ήταν ένας καλός νόμος για τις ποσοστώσεις. Έγινα 62 ετών, παλεύω εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το θέμα στη χώρα μου και παγκοσμίω. Έχω βαρεθεί τους στόχους. Δεν λειτουργούν. Χρειάζεται, όπως είπε και η κυρία Τσίμερμαν, κάποια στιγμή η καλή θέληση δεν αρκεί, χρειάζεται νομοθεσία. Ποια είναι λοιπόν η ορθή νομοθεσία. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν και θα το μοιραστώ αυτό με την Επιτροπή σας και είναι σημαντικό ε, για να το βάλετε στη συστάση σας εάν πάτε προς ποσοστός. Χρειάζεται ένα σχέδιο εφαρμογής. Κάποιες από τις νομοθεσίες δεν είχαν τέτοιο σχέδιο. Πέρασαν τον νόμο και δεν ήξεραν τι να κάνουν μετά η, στην Νορβηγία λειτουργήσε γιατί είχαν ένα σχέδιο εφαρμογής για το πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δεύτερον, πρέπει να δοθούν οι πόροι. Δεν μπορούμε να περάσουμε ένα νόμο χωρίς χρήματα. Πρέπει να έχει κονδύλια για, που να πάνε στο Υπουργείο το επιφορτισμένο με αυτή τη δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν, όπως ακούστηκε, κυρώσεις, ποινικά μέτρα Χωρίς αυτό οποιαδήποτε νομοθεσία δεν έχει νόημα, κανείς δεν ακολουθήσει το νόμο γιατί είναι ωραίος. Ο λόγος για τον οποίο πέρασε ο νόμος στην Ορβηγία ήταν πως το πέρασαν τρεις κυβερνήσεις, από συντηρητική μέχρι προοδευτική. Οπότε πρέπει να υπάρχει καλή θέληση από όλους τους εταίρους ενός σχηματισμού για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο ενός συνασπισμού. Κατόπιν προθεσμίες τις οποίες πρέπει να τηρήσουν όλοι και είμαι περίεργη για το τι θα γίνει στην Γαλλία όταν αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια βάση δεδομένων ικανών γυναικών. Ίσως να μην τη χρησιμοποιήσουν η εταιρεία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός γυναικών που θα είναι έτοιμες και τέλος εκπαίδευση ανδρών και γυναικών σε ζητήματα εταιρική διακυβέρνηση. Γιατί οι εταιρείε ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν μεγάλε προκλήσει και είναι σημαντικό όπως βγαίνουμε από αυτή την κρίση να δούμε όχι μόνο ποιες είναι οι ρυθμιστικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αλλά στο ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές. Ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείε αναπτύσσονται σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχουν επιρροή και αντίκτυπο στους εργαζόμενους παντού, στις οικονομίες, στο περιβάλλον, εκεί όπου δραστηριοποιούνται. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να έχουν λόγο στα ΔΣ που επιβλέπουν αυτές τις εταιρείε. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστούμε κυρία Νατιβιδά. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην άλλη Αμερικανίδα προσκεκλημένη μας, την κυρία Ελισάβετ Μπένχαμ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας επιχειρηματίνων. Σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσω ευχαριστώντας την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών για την πρόσκλησή της. Είναι για μας μεγάλη τιμή που μιλούμε σήμερα μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος της οργάνωσής μας και μάλιστα για θέμα που το θεωρούμε πολύ σημαντικό για την προώθηση των γυναικών στην οικονομία και στη λήψη αποφάσεων. Η οργάνωσή μας είναι μίκη όμικρον και σήμερα γιορτάζει την 80η της επέτειο. Έχει δε μέλη σε 96 χώρες, πάνω από 30.000 μέλη και με μεγάλη χαρά αποτελώ την 21η της πρόεδρο. Έχει ρόλο στο και για πάνω από 60 χρόνια προωθεί θέματα γυναικών, ιδιαίτερα την ισότητα των φύλων. Τελευταία έχουν σημειωθεί αρκετές νίκες για τις γυναίκες, αλλά ο τόπος εργασίας παραμένει ανδρικός. Αν και έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές, οι γυναίκες δυστυχώς ζουν τεράστια ανισότητα. Η τελευταία μελέτη McKinsey Global δείχνει ότι η πλειοψηφία των διευθυντικών στέλεχων θεωρεί ότι η ποικιλομορφία των φύλων σε διευθυντικές θέσεις οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα αλλά δεν ε, υπάρχουν οι ανάλογοι διορισμοί. Φαίνεται ότι έχει αυξηθεί μεν το μερίδιο των γυναικών παρά την κρίση, αλλά παρόλα αυτά οι εταιρείε μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ανώτατες θέσεις. Και αυτό δεν είναι εκπληκτικό, διότι η μελέτη δείχνει ότι δεν είναι μεγάλη προτεραιότητα η ισότητα των φύλων για τις εταιρείε και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην πολιτική που ακολουθούν για τα φύλλα. Λόγω αυτών των δύο παραγόντων τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το περισσότερο είναι καλύτερο, δηλαδή ότι σε εταιρείες όπου υπάρχει περισσότερη ισότητα των φύλων, εκεί τα διευθυντικά στελέχη λένε ότι και η ηγεσία της εταιρείας είναι η πιο διαφοροποιημένη. Οι εταιρείε που έχουν μεγαλύτερη ισότητα των φύλων παρουσιάζουν 32% διαφορά μεταξύ του μεριδίου των γυναικών που αντιπροσωπεύουν πάνω από 15% των θέσεων τύπου Γ και Άνω. Και άνω. Ο αριθμός στήριξης από μήκη όμικρον είναι άλλο σημαντικός παράγον που επηρεάζει τα αποτελέσματα μιας εταιρεία και γι' αυτό φαίνεται ότι λίγες μόνο εταιρείε έχουν στα ανώτατα συμβούλια τους προγράμματα για την ισότητα των φύλων. Οι διαφορές που αναφέρουν τα διευθυντικά στελέχη στις περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν ότι όλες οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση και ως προς τα φύλλα και επομένως και τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Είναι μεγάλη βέβαια προτεραιότητα η ισότητα, αλλά το θέμα είναι και πόσες γυναίκες υπάρχουν στις ανώτατες θέσεις. Σε εταιρείε όπου αυτό είναι προτεραιότητα, 80% των ερωτωμένων λένε ότι πολύ λίγες γυναίκες είναι στις υψηλότατες θέσεις και μόνο 60%, 64% των εταιριών τις θεωρούν προτεραιότητα. Επίσης υπάρχουν και γεωγραφικές διαφορές. Οι ερωτώμενοι στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και σε αναπτυσσόμενες αγορές λένε ότι η διαφοροποίηση των φύλων, η ισότητα μάλλον των φύλων είναι βασικό θέμα για την εταιρεία τους 35 και 34% δυστυχώς από τις υπόλοιπε υπόλοιπες περιοχές. Στη Λατινική Αμερική μόνο 21% των ερωτωμένων θεωρούν ότι οι εταιρείε τους συμπεριλαμβάνουν ως προτεραιότητα την ισότητα των φύλων και 27% στην Ευρώπη και 28% στη Βόρεια Αμερική. Κατά τα ταξίδια μου σε ολόκληρο τον κόσμο σε διασκέψεις, μεταξύ των οποίων και το δίκτυο γυναικών ΑΠΕΚ στην Ιαπωνία, όλα δείχνουν το ίδιο πράγμα και συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις δεν αντιδρούν αρκετά γρήγορα ενώ οι επιτυχίες δείχνουν τι χρειάζεται. Αφού χρειάζεται να υπάρξει μια κρίσιμη μάζα γυναικών που να αλλάξει τα πράγματα και μια κρίσιμη μάζα γυναικών σε ανώτατες θέσεις σημαίνει και την αποδοχή της διαφοράς. Οι αποφάσεις που αφορούν την προώθηση των γυναικών και την προαγωγή των γυναικών είναι επίσης σημαντικό θέμα. Οι ποσοστώσεις μας έχουν δείξει ότι έχουν αποτέλεσμα και τις θεωρούμε ως σημαντικό μέσον για να αρχίσει η αλλαγή που χρειάζεται τόσο πολύ και να κινηθούν οι γυναίκες προς τα επάνω στις διευθυντικές θέσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι η εξισορρόπηση των φύλων να αποτελέσει τη βάση της λειτουργίας της εταιρείας ώστε περισσότερες γυναίκες ανώτατα στελέχη να διορίζονται και να έχουν έτσι και το κίνητρο να ζητήσουν τέτοιες θέσεις. Το θέμα είναι το εξής. Μόλις υπάρχουν τρία μέλη γυναίκες του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζουν να φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα. Ποιο είναι όμως το κύριο θέμα, ο αριθμός ή η διευκόλυνση της λήψης, της κατάληψης των θέσεων στην Αυστραλία θεωρήθηκε από το χρηματιστήριο προτεραιότητα η ισότητα των φύλων και ζήτησε από εταιρείε να εφαρμόσουν και να δημοσιεύσουν διάφορα προγράμματα που να καθορίζουν περισσότερη ισότητα των φύλων από του χρόνου ήδη αναμένεται οι εταιρείε να δημοσιεύσουν αν έχουν πετύχει τους στόχους αυτούς και να δημοσιεύσουν επίσης το ποσοστό γυναικών σε ανώτατες θέσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπολογίζει ότι ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι 18,7% εκατομμύρια γυναικών έχουν πέσει στην ανεργία. Οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό ε, από τους άνδρες για την ίδια εργασία, κερδίζοντας ένα 70-90% των μισθών των ανδρών. Ενώ αυτό το μισθολογικό χάσμα έχει μειωθεί από το 2000 έως το 2007, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τροχοπέδης η BPW International προβάλλει μία εκστρατεία ίσης ε, μισθοδοσίας για να μειώσει αυτό το χάσμα. Αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μία σειρά κατευθυντηρίων γραμμών έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να αναλάβουν δυναμικό ρόλο. Θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη την κοινή πρωτοβουλία UNIFAM και UN Global Compact Women's Empowerment Principles. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι μία μεγάλη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του παγκοσμίου δικτύου. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε τον πραγματικό ρόλο τους στις γυναίκες στο, στην παγκόσμια αγορά και στην αγορά εργασίας. Αυτό αφορά ηγετικές θέσεις, ίσες ευκαιρίες και μη διάκριση έτσι ώστε να έχουν την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση να ε, βοηθήσουμε δηλαδή και τις γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο. Η αρχή παριθμών 7 ενθαρρύνει τις γυναίκες να ε, ορίσουν ορόσημα και διαφανείς διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί μιλώντας για στοιχεία, δίνοντας στοιχεία που δεν βασίζονται στο φύλλο. Με βάση τη συμμετοχή της BPW International, φέτος το Μάρτιο, αυτές οι αρχές πλαισιώνονται από συγκεκριμένες πρακτικές, από επιχειρήσεις διατομιακά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε πραγματοποιήσιμους στόχους. Υπάρχει μία σειρά νέων κανόνων έτσι ώστε να φτάσουμε στην εξισορρόπηση τη μισθολογική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θεωρούμε ότι τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να έχουμε μετρήσιμους στόχους για να μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει μια σωστή πολιτική. Ε, έχουμε έρθει σε επαφή με θηγατρικές όλο τον κόσμο, με μέλη σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε να συνεργαστούμε και με κυβερνητικούς φορείς και με επιχειρήσεις για να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που ε, δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες στις γυναίκες και μέσω διαδικτύου. Θεωρούμε ότι η δήλωση του Ιουνίου στην διάσκεψη κορυφής των ε, επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη ε, όρισε αυτούς τους στόχους έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των γυναικών να χρησιμοποιήσουν αυτές τις αρχές. Πάνω από 100 ε, διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ε, υπογράψει αυτή τη δήλωση θεωρώντας ότι η ισότητα είναι το σωστό και το πιο ε, έξυπνο που θα πρέπει να γίνει. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μεγάλη και σημαντική εργασία έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική στήριξη των γυναικών στην παγκόσμια αγορά, αγορά εργασίας και την κοινότητα θα πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας δηλαδή για την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και για τις γυναίκες και από τις γυναίκες. Χωρίς ε, να ε, μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε αυτούς τους στόχους, δεν θα ενισχύσουμε ούτε το ρόλο της γυναίκας. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα Μπανκιμούν, ο οποίος στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας μίλησε για αυτά τα προγράμματα. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από τους παγκόσμιους ηγέτες και τους, ε, τον επιχειρηματικό κόσμο για να επιταχύνουμε την πρόοδο. Ποτέ δεν είχαμε δει μια τέτοια σύγκληση των διεθνών εμπλεκόμενων φορέων για τη συμμετοχή των γυναικών σε, όλους, σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε επαρκώς αυτό το δυναμικό. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να έχει αυτή η επιτυχία και να ορίσουμε και τις μεθόδους και τα μέσα. Δεν θα πρέπει να γίνει το αντίστροφο. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση στασιμότητας. Θα πρέπει να υπάρχει βιώσιμη δέσμευση σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα. Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι το ίδιο. Αποτελούν και ορίζουν τις ε, ίδιες αρχές. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο και η BPW θα συνεχίσει με επιμέλεια αυτή την εργασία έτσι ώστε αυτό, αυτό το πλαίσιο να αποτελέσει πραγματικότητα. Εάν η, η ισότητα είναι ένα δικαίωμα που απορρέει από τη γέννηση του ανθρώπου, γιατί να δεχτούμε οτιδήποτε λιγότερο. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπένχαμ, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Καθώς και όλους όσους έλαβαν το λόγο στο πάνελ αυτό. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη, στους βουλευτάς. για να κάνουν σχόλια. Λοιπόν, Ας δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Ιντακής που αντικαθιστά την κυρία Τσεσκόβα που είναι σκιώδης εισηγήτρια εξ ονόματος των συνδυρητικών. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω όπως είπατε και εσείς εξ ονόματος της συναδέλφους μου κυρίας Ανδρίας Τσεσκόβα που καθυστέρησε στις αεροπορικές. Η δουλειά μου είναι πολύ εύκολη, θα σας διαβάσω το έγγραφό της. Θα μπορούσα να κάνω και δικά μου σχόλια βέβαια, αλλά να θα το διαβάσω. Λοιπόν, αρχίζω πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε υπεύθυνε θέσεις. Επίσης όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι εργοδότες πρέπει να έχουν ελαστικότητα ως προς το ποιον διορίζουν. Στην τσεχική δημοκρατία το μερίδιο των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις είναι 9,5%. Αυτό πλησιάζει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 11%. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο αριθμός είναι ακόμη πολύ μικρός. Η κύρια όμως ανησυχία είναι ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν φραγμούς από τη στιγμή που μπαίνουν σε μια υπεύθυνη θέση. Ας πούμε αν αποφασίσουν να αρχίσουν να κάνουν μια οικογένεια, να δημιουργήσουν μια οικογένεια, πρέπει να τους δοθούν οι κατάλληλες συνθήκε εργασίας δηλαδή ευέλικτο ωράριο εργασίας, παιδικούς σταθμούς με ευέλικτο ωράριο. Όπα. Ένας άντρας εδώ πέρα ήρθε να μας σώσει. Ευελιξία για να δουλέψουν στο σπίτι, εταιρική παιδική σταθμή, κατάλληλοι χώροι που τους επιτρέπουν να θυλάζουν τα νεογέννητα. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι οι γυναίκες να μην αναγκάζονται να παίρνουν υποχρεωτική άδεια μητρότητας. Σημαντικό είναι να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την επιλογή. Δεν πρέπει μόνο να λέμε ότι έχουμε πολιτικές ε, προτεραιότητες, πρέπει να αλλάξουμε και τις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων. Επίσης, σημαντική είναι η κάλυψη από τα ΜΜΕ για να αυξηθούν οι γυναίκες ε, στη λήψη αποφάσεων μέσω της προβολής π.χ. γυναικείων προτύπων. Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις για να αυξηθούν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις επίσης θα πρέπει να αποφευχθεί. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ένας, έναν από τους λόγους χαμηλής εκπροσώπησης γυναικών σε ηγετικές θέσεις που οφείλεται στην απόφαση των ιδίων των γυναικών. Πολλές γυναίκες επιλέγουν να έχουν οικογένεια και όχι καριέρα. Μπορεί να επιλέξουν να σταματήσουν τις καριέρες τους και να τις συνεχίσουν αργότερα όταν έχουν φύγει τα παιδιά από το σπίτι όπως είπα και νωρίτερα, ευκαιρίες και ευελιξία είναι αυτό το οποίο έχει σημασία για να διαμορφώσουν την φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός σπιτιού. Και νομίζω πως θα μείνω στα σχόλια της ε, Άντριας και θα ρωτήσω τα δικά μου για την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Um, Τώρα θα δώσουμε το λόγο στη, στην ιστόν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Ντανιέλα Μπανκέ έχει το λόγο που είναι επικεφαλής ομάδα, της ομάδας μονάδας συγγνώμη, μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακρόαση αυτή για τις γυναίκες σε ηγετικέ θέσει, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να είμαι σύντομη γιατί ήταν μεγάλο το απόγευμα, ακούστηκαν ήδη ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και Αυτά τα οποία άκουσα νομίζω τόνισαν τα σημαντικότερα σημεία. Αυτό το οποίο, στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι το πώς βλέπει η Κομισιόν το θέμα των γυναικών στην λήψη αποφάσεων και τι σκοπεύει να κάνει για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματα στον τομέα αυτών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο νούμερα για το πώς ε, το πού βρίσκονται οι γυναίκες σήμερα στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, σήμερα στην Ευρώπη κατά μέσο όρο έχουμε ένα στα δέκα μέλη στα δέλτα σίγμα μεγάλων εισηγμένων εταιριών. Γύρω στο 10% μιλάω για εποπτικά συμβούλια, όπως είπα, μεγάλων εισηγμένων εταιριών είναι γυναίκες και μόνο 3% προέδρων ΔΣ είναι γυναίκες. Οπότε βλέπετε τα νούμερα είναι άσχημα και αυτό το οποίο είναι πιο ανησυχητικό από τα νούμερα της σημερινής κατάστασης είναι πως η τάση δεν βλέπουμε κάποια τάση βελτίωσης της κατάστασης. Βλέπουμε πως τα νούμερα παραμένουν σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια και άρα θεωρούμε πως είναι ενισχυτικό το φαινόμενο και επίμονο αν θέλετε. Και αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μία παρένθεση, η Κομισιόν βγάζει αυτές τις εκθέσεις για τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων εδώ και κάτι χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μία βάση δεδομένων που καλύπτει και τις πολιτικές και τις οικονομικές λήψη αποφάσεων αναφέρθηκε ήδη η βάση δεδομένων γιατί πριν από κάτι χρόνια διαπιστώσαμε ότι γίνεται πολλής λόγος για τις γυναίκες και τα κενά και τα λοιπά, αλλά κανείς δεν έχει νούμερα. Οπότε κάναμε αυτή τη βάση δεδομένων, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας και δημοσιεύουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εκθέσεις αυτές. Έχουμε φέρει και κάποιες μαζί μας σήμερα, αν ενδιαφέρεστε. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν ποια είναι τα γεγονότα. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση, τα νούμερα ε, δεν είναι θετικά. Δεν υπάρχει κάποια τάση βελτίωσης της κατάστασης, οπότε η Κομισιόν θεωρεί πως οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες ε, στις οποίες θα εστιάσει στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Κομισιόν υιοθέτησε την ε, μεσοπρόθεσμη στρατηγική της για τα επόμενα πέντε χρόνια για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και όπως σας είπα μία από τις πέντε προτεραιότητες του νέου προγράμματος Κομισιόν είναι οι γυναίκες στη λήψη για να σας δώσω να καταλάβετε σε τι επίπεδο το βάζουμε, οι άλλες τέσσερις ε, προτεραιότητες είναι η οικονομική ανεξαρτησία, η βία κατά των γυναικών, το κενό στις πληρωμές και η ισότητα στις εξωτερικές σχέσεις. Οπότε για μας η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό τον τομέα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ο προφανής λόγος της ισότητας, της δικαιοσύνης, πρέπει οι γυναίκες να εκπροσωπούνται εξίσου και σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας και δεύτερον θεωρούμε πως είναι και σωστό επιχειρηματικά για περισσότερες γυναίκες ε, να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία των επιχειρήσεων συμφωνώ με κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν θεωρούμε πως είναι σωστό επιχειρηματικά Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν μια θετική σχέση μεταξύ της παρουσίας γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και της απόδοσης των επιχειρήσεων. Αν και νομίζω πως α, ακόμα αξίζει να το διερευνήσουμε, να ερευνήσουμε καλύτερα αυτόν τον τομέα για να ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας για το σχετισμό αυτών αλλά βλέπουμε και αναφέρθηκε αυτό πως και οι γυναίκες και οι άντρες στη διοίκηση των ευρωπαϊκών εταιριών θεωρούν πως η ισορροπή συμμετοχή είναι μια οικονομική αναγκαιότητα για τις εταιρείες σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχουν καλοί λόγοι για να επιτύχουμε πρόοδο εδώ πέρα και η κυρία Ρέντινγκ, η επιτροπός μας που τα ανακοίνωσε αυτά και στο Κοινοβούλιο πρόσφατα σε μια ανταλλαγή απόψεων που είχε είπε πως σκοπεύει να προβεί σε απευθείας διάλογο και επαφές με τους επικεφαλείς ευρωπαϊκών εταιριών θέλει να μπει σε ένα τέτοιο διάλογο για να συζητήσει μαζί τους τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και ο διάλογος αυτός θα γίνει για πρώτη φορά την άνοιξη του επόμενου έτους με βάση ένα έγγραφο το οποίο θα συντάξει η Κομισιόν στο οποίο θα έκτιμα την κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση των γυναικών σήμερα στην Ευρώπη, στις επιχειρήσεις και θέλει επίσης η Κομισιόν στο έγγραφο αυτό να εξετάσει τι, ποια είναι τα πιθανά μέτρα για να γεφυρωθεί το κενό και να διασφαλίσουμε πως υπάρξει βελτίωση στον τομέα αυτών. Αυτά μπορεί να είναι μέτρα εθελοντικά που μπορεί να βοηθήσει η κυβέρνηση, μπορεί να είναι μέτρα μη νομοθετικά αλλά και νομοθετικά. Οπότε θέλουμε να θέσουμε επιτάπητος ε, τις δυνατότητες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και με βάση αυτόν τον απολογισμό που θα κάνουμε η Κομισιόν θα επιζητήσει διάλογο με τις μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης για να δούμε τι είναι διατεθειμένες να κάνουν. Και βεβαίως αυτό το οποίο προτιμάμε είναι οι εταιρείες να δεσμευτούν εθελοντικά για να βελτιώσουν την κατάσταση. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να δίνουμε αναφορά τακτικά για τις εξελίξεις και ελπίζω την πρόοδο. Θα συνεχίσουμε και κάτι που ξεκίνησε στο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε δηλαδή αυτό το δίκτυο γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Ξεκίνησε πριν από κάτι χρόνια από την Κομισιόν και χαίρομαι που κάποιες ε, στο βήμα αυτό το έχουν ακούσει είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκό και προσπαθούμε εκεί να ανταλλάσσουμε ορθές πρακτικές και να δούμε ποια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν περισσότερες γυναίκες να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα στις επιχειρήσεις και στην πολιτική. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή η προσπάθεια δικτύωσης και τέλος νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ε, τα μέτρα για την αύξηση του αριθμού γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις νομίζω πως δεν θα επιτύχουν μεμονωμένα. Πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας πιο συνολικής προσέγγισης μέρος πολιτικών που θα στοχεύουν στην διεύρυνση του αριθμού των γυναικών που είναι ικανές να είναι μέλη ΔΣ. Πρέπει να διευρυνθεί αυτός ο αριθμός. Παραδείγματο χάρη με το να είναι πιο εύκολο να ε, συμβιβάσει κανείς τις υποχρεώσεις της δουλειάς και της οικογένειας αλλά και με το να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να επιλέξουν ε, σπουδές που οδηγούν σε αυτές τις θέσεις. Πρέπει δηλαδή να διευρυνθεί ο αριθμός των γυναικών που είναι διατεθειμένες να είναι μέλη ε, ΔΣ. Αυτό θα γίνει και με το να ενθαρρύνουμε άντρες να τις βοηθήσουν ως συνάδελφοι παραδείγματο χάρη στις επιχειρήσεις αλλά και ως σύντροφοι με το να ε, τις βοηθήσουν το... Η επόμενη σημαντική λοιπόν ημερομηνία είναι η Άνοιξη, η οποία έρχεται όταν θα συναντηθεί η Επίτροπος με Ευρωπαίους Διευθύνοντες Συμβούλους μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεχίσουμε με τα συνοδευτικά μέτρα, τις πολιτικές που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπανκέ, σας ευχαριστούμε πολύ διότι μας ε, είπατε πώς ε, αντιμετωπίζει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε διότι αυτό το θέμα είναι μία προτεραιότητα για σας και για την Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ. Τώρα τα μέλη βουλευτές μπορούν να λάβουν το λόγο. Έχω έναν κατάλογο ομιλητών. Η κυρία Ματέρα είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις των εισηγητριών σε αυτή την ε, ακρόαση και αυτό που έχει σημασία είναι να ε, δούμε ε, πώς, είχε, πώς είχαν παρεμβάσεις και ιδιαίτερα στις κυρίας Νατιβιδάτ που ε, εκπροσώπησε, εκπροσω... όπου εκπροσωπήθηκαν όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως είναι πρόδειλο ότι η Νορβηγία είναι το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς φτάνουμε στους απότερους στόχους. Να δούμε πώς θα ορίσουμε ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. Και θα πρέπει να ληφθεί η υπόψη και η κατάσταση της, ε, στη δική μας χώρα. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα 3% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να σπάσουν αυτό το φράγμα. Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να κατέχουν διευθυντικές θέσεις, θέσεις στα διοικητικά συμβούλια. Και θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση δεν νομίζετε ότι ε, αυτό το ζήτημα όπως το προωθούμε αποτελεί μία τροχοπέδη. Δηλαδή φαίνεται ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε για να φτάσουμε σε συγκεκριμένους ε, στόχους. Γιατί ε, στη Νορβηγία η ισχύει αρχή των Golden Skirts. Θα πρέπει Επίσης να δούμε ποιες είναι οι κυρώσεις που επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση τη στιγμή που δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των ποσοστώσεων. Ευχαριστούμε. Κυρία Ματέρα. Η κυρία Λούλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν με συγχωρείτε που ήρθα καθυστερημένη, είχα άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά με βάση αυτά που άκουσα θα ήθελα να προσέξουμε ορισμένες πολύ ορισμένα πολύ γενικά αιτήματα, παραδείγματος χάρη για τις ποσοστώσεις στις διευθυντικές θέσεις των μεγάλων εταιριών γιατί μπορεί έτσι να παραγνωρίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στις 27 χώρες μέλη ως προς το εταιρικό δίκαιο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και αν ζητήσουμε ποσόστοση 40% πρέπει να δούμε και πού θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Στο εταιρικό δίκαιο των λατινικών, για να το πω έτσι, χωρών Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει ένα Aufsichtsrat, εποπτικό συνέδριο, το οποίο είναι άλλο πράγμα από το διοικητικό συμβούλιο στο εταιρικό δίκαιο του ρωμαϊκού δικαίου. Επομένως, αν ζητήσουμε 40% για το Aufsichtsrat στη Γερμανία, Γίνεται, εξάλλου υπάρχει και συνδιεύθυνση στο Aufsichtsrat. Αν ζητήσουμε όμως 40% στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας στο εταιρικό δίκαιο του Ρωμαϊκού Δικαίου, τότε άλλο πράγμα, για άλλο πράγμα μιλάμε και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε τις διαφορές ως προς το εταιρικό δίκαιο των χωρών μελών και τι σημαίνουν τα αιτήματά μας διότι δεν έχουμε ποσόστοση στη χώρα μας για τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών Action Gesellschaft στα γερμανικά, νόημη εταιρεία. Αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά, υπάρχει και η συνδιαχείριση, είπα, στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε εκπροσώπους των συνδικάτων που συμμετέχουν στο Aufsichtsrat. Δεν είναι το ίδιο καθοριστικά όπως τα διοικητικά συμβούλια. Ενώ σε εμά είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα όταν κάνουμε, διατυπώνουμε αιτήματα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Ότι δηλαδή το εταιρικό δίκαιο διαφέρει από χώρα σε χώρα και ζητάμε πολύ περισσότερα σε μια χώρα στην πράξη από ό,τι στην άλλη ε, με την ίδια διατύπωση ανάλογα με το εταιρικό δίκαιο. Κάτι άλλο τώρα. Και εγώ πριν από πάνω με, από 20 χρόνια είχα ζητήσει να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες θετικές δράσεις για τις γυναίκες στη χώρα μου στο Λουξεμβούργο σε μια τράπεζα. Είχα ζητήσει από τον Σύλλογο Τραπεζιτών και Τραπεζών αν συμφωνεί να γίνει κάτι τέτοιο σε όλες τις τράπεζες είχαν πει βεβαίως, βεβαίως αλλά δεν βρίσκουμε γυναίκες που να είναι διατεθειμένες να αναλάβουν τέτοιες διευθυντικές θέσεις και διαπίστωσα και εγώ ότι όλες οι γυναίκες που είχαν κάποια σταδιοδρομ... τραπεζική στρατιοδρομία είτε ήταν ανήπαντρες είτε ήταν χωρισμένες χωρίς παιδιά καμία όμως δεν είχε κανονική οικογένεια με παιδιά μάλιστα μικρή ηλικία. και γιατί αυτό διότι βάσει της νοοτροπίας που δυστυχώς δεν έχει αλλάξει της κυρίαρχης νοοτροπίας η κατανομή των ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ζεύγη δεν είναι ιδεώδης. Σε ένα διοικητικό συμβούλιο τραπέζης ή αν είστε διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας και σας πει η Λουξεμβουργική Τράπεζα αύριο να είστε στη Σιγκαπούρη γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα τηλεφωνάει ο διευθυντής στη γυναίκα του και λέει ετοίμασε τη βαλίτσα μου ενώ η γυναίκα τι θα έκαμνε αναρωτιέται σε τέτοια περίπτωση τι θα γίνουν τα παιδιά, ποιος θα ετοιμάσει το φαΐ. Πολλές, πολλά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν οι άντρες και γι' αυτό διστάζει να δεχτεί τέτοιες θέσεις. Έτσι μου είπανε και εγώ αυτό διαπίστωσα, το ξέρω και εγώ. Δεν έχω μεν άντρα και παιδιά, Άρα για μένα είναι εύκολο, μπορώ να πάω αύριο στη Σιγκαπούρη, γι' αυτό έρχομαι και κάθε μέρα στις Βρυξέλλες εδώ. Αν είχα άντρα και παιδιά θα με είχε διώξει από πολύ καιρό. Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν διαφορές και ότι δυστυχώς οι γυναίκες συνήθως έχουν να σκεφτούν την οικογένειά τους πιο πολύ από ότι οι άντρες. Δεν ξέρω οι νέες αν το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω δεν άλλαξαν πολύ τα πράγματα δυστυχώς. Λοιπόν, έγινε λόγος και για τις διαφορές των μισθών. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε με τις στατιστικές, με τα στατιστικά στοιχεία. Πριν από μερικά χρόνια ακούστηκαν στατιστικά στοιχεία για τις μυθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη βιομηχανία σε επίπεδο εργατών όχι στελεχών και η χώρα μου έχει ψηλούς μισθούς νομίζω ότι είναι μάλιστα η υψηλότερη των, στην Ευρώπη στην Ένωση και βρέθηκε στον πάτο γιατί εκεί υπήρχαν οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ εργατών και εργατριών ως προς τους μισθούς. Γιατί. Γιατί αυτό εξαρτάται από τη δομή της βιομηχανίας. Η χαλιβουργία κυριαρχούσε τότε και στη χαλιβουργία ή στα ορυχεία δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες τουλάχιστον σε ποιοτικέ θέσεις. Μερικές χαμάλισες υπάρχουν στη Χαλιβουργία, αλλά δεν υπάρχουν γυναίκες που να εργάζονται στις υψικαμίνους ή κάτω στα ορυχεία και οι ειδικευμένοι εργάτες στη Χαλιβουργία ευτυχώς πληρώνονται παραπάνω από ό,τι οι χαμάλιδες ευτυχώς, ή της καθαρίστρης, του καθαριστάς. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όταν ερμηνεύουμε στατιστικά στοιχεία για μέσους όρους που να καλύπτουν ολόκληρη χώρα. Εξαρτάται, πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Να γνωρίζουμε τη δομή της οικονομίας μιας χώρας. Δεν αρνούμε δεν αρνούμε ότι υπάρχουν διαφορές. Και εγώ είμαι θύμα των διαφορών αυτών, των μισθολογικών διαφορών, διότι άρχισα να εργάζομαι όταν ακόμη ήταν νομικά δυνατόν να δίνονται χαμηλότεροι μισθοί στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Και η δική μου γενιά έχει συντάξεις, οι γυναίκες έχουν συντάξεις πολύ υψηλότερες από τον αντρών. Γιατί, γιατί χαμηλότερες μάλλον από τον αντρών εννοεί η ομιλήτρια, γιατί υπήρχαν διαφορετικοί μισθοί. Δεν κατάφερα βέβαια ποτέ να πάρω τη συνταξή μου, αλλά τέλος ε, πρέπει να προσέχουμε. Εγώ τολμώ και το λέω, γιατί δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι δεν μιλάω υπέρ των γυναικών, το κάνω εδώ και 50 χρόνια περίπου. Εξάλλου όταν έγινα βουλευτή πριν από 45 χρόνια δεν υπήρχαν τουαλέτες γυναικών. Χαμάλισες και καθαρίστριες μπορεί να υπήρχαν αλλά δεν τις έβλεπα Δεν μπορείτε λοιπόν να μου πείτε ότι δεν μιλάω υπέρ των γυναικών, αλλά και είμαι ακόμη πρόεδρος μιας γυναικείας οργάνωσης και μέχρι πριν από ένα χρόνο ήμουν και πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Γυναικών στη χώρα μου. Δεν είμαι υποπτή λοιπόν, αλλά θέλω να είμαστε ρεαλίστριες. Εγώ κατάφερα να πετύχω πολλά πράγματα για τις γυναίκες στη χώρα μου επειδή ήμουν ρεαλίστρια. Και με μαξιμαλιστικά αιτήματα δεν καταλήγουμε πουθενά. Πρέπει να είμαστε ρεαλίστριες και αντικειμενικές. Και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Αν όμως μερικοί λένε ή μερικές ότι οι μισθολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών υπάρχουν, πράγμα που είναι σωστό. Από το 75 όμως διαθέτουμε μια πολύ καλή οδηγία για την για τους ίσους μισθούς, για την ισότητα των μισθών και στη χώρα μου, εγώ κατάφερα πάρα πολλά πράγματα με βάση αυτή την οδηγία που ισχύει ακόμη και είναι ακόμη σωστή. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να έχει κανείς το θάρρος, αν καταλαβαίνει τα πράγματα, να ζητήσει την εφαρμογή του δικαίου. Ένα παράδειγμα, σε μια κοινότητα είχα κάνει μια δίκη γιατί οι καθαρίστριες πληρώνονταν λιγότερο από τους καθαριστάς και την κερδίσαμε τη δίκη. Ήταν καμιά εικοσαριά καθαρίστριες που πληρώθηκαν και εκ των υστέρων 20 εκατομμύρια λουξεμβουργικά φράγκα τότε η κοινότητα βέβαια ήταν έξαλλη κατά εμού, αλλά αναγκάστηκε να πληρώσει. Και για να μην μακρηγορήσω θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις είχαμε ανάλογες επιτυχίες γιατί όταν κανείς τολμήσει να φτάσει μέχρι τα δικαστήρια και να απαιτήσει την επιβολή του δικαίου πετυχαίνει. Το έκανα και όταν ίσχυε στο Λουξεμβούργο με βάση αυτή την οδηγία η επιχορήγηση αρχηγού οικογενείας και για γυναίκες και αυτό είχε κοστίσει την εποχή εκείνη το 70 700 εκατομμύρια στο κράτος του Λουξεμβούργου, 700 εκατομμύρια φράγκα για πληρωμές γυναικών εκ των υστέρων που δεν είχαν πάρει επίδομα αρχηγού οικογενείας. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αναδρομικά. Να σας πω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας βοήθησε πάρα πολύ αλλά πρέπει να έχει κανείς το θάρρος να την εφαρμόσει και να ζητήσει την εφαρμογή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λούλιν. Είμαστε πεπισμένοι και πεπισμένες ότι η κυρία Λούλιν έχει το θάρρος να αναλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα, διότι είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι κάποια μέρα οι γυναίκες θα είναι πραγματικά ίσες έναντι των ανδρών και θα αναλαμβάνουν τα ίδια καθήκοντα και ίσως αντιστραφούν και οι ρόλοι. Θα ήθελα τα μέλη του πάνελ τώρα να αντιδράσουν. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εισηγήτριες για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Όλοι μιλάμε για ίση εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην επιχείρηση. Ναι, μιλάμε για, μια, ε, για έναν ίσο επιμερισμό ευθυνών. Φαίνεται το σύστημα των ποσοστώσεων είναι λειτουργικό. Νομίζω όμως ότι πριν από αυτό θα πρέπει να εργαστούμε στο τομέα της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, διότι και οι ε, άντρες θα πρέπει να είναι κοινωνοί του θέματος. Δυστυχώς οι άνδρες είναι μεγάλοι απόντες και από αυτή την αίθουσα και νομίζω ότι θα πρέπει άνδρες και γυναίκες να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση, να αλλάξουμε τα στερεότυπα, να συνεκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ε, μία αμφίδρομη πορεία, μία αμοιβαιότητα. Να υπάρχει αυτή η ισορροπημένη εκπροσώπηση. Στην Ισπανία έχουμε το νόμο περί σε ορισμένες περιφέρειες. Γι' αυτό, ε, για παράδειγμα, θα πρέπει να λέγεται ο ή στους εκλογικούς καταλόγους και να υπάρχει ίσως αριθμός υποψηφίων Αυτό είναι ζήτημα αρχής. Δηλαδή είχαμε να κάνουμε, είχαμε να κάνουμε ένα νόμο ποσοστώσεων όπου υπήρχε μεν ίση εκπροσώπηση, αλλά οι γυναίκες ήταν τα τελευταία ονόματα της λίστας. Νομίζω τέλος πάντων ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της εκπαίδευσης. Ως προς τη γυναίκα επιχειρηματία, Νομίζω ότι υπάρχει, εθνική, ε, υπάρχει σωστή αντιμετώπιση, αλλά πολλές φορές οι γυναίκες δουλεύονται για κάποιον τρίτο, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις υπεργολαβίας και ούτω καθεξής και η γυναίκα δεν μπορεί να έχει τις 16 εβδομάδες όταν εργάζεται σε μια μικρή επιχείρηση και θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το φράγμα και να μας απασχολήσει το θέμα του πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε μία γυναίκα επιχειρηματία η οποία χτίζει μία επιχείρηση. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη ότι και τα ε, ε, παιδιά και τα, ας πούμε, και τα παιδιά μας μπορούν να συμμετέχουν σε, σε ε, διάφορες επιχειρήσεις, στα διοικητικά συμβούλια, αλλά ε, παραδείγματος χάρη κάποιος που δουλεύει στις Βαλιαρίδες νήσους ίσως θα πρέπει να μεταβεί ξαφνικά στην Αργεντινή για να συνάψει ένα συμβόλαιο. Ε, για μας είναι εύκολο, διότι είμαστε ευρωβουλευτές, αλλά ας λάβουμε υπόψη ότι και στον τομέα των υπηρεσιών δεν ισχύει πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ορισμένες υπηρεσίες. Εμείς μπορούμε να καταβάλουμε το, αντίτυπο, το αντίτιμο με συγχωρείτε ορισμένων υπηρεσιών, αλλά ε, γυναίκες χαμηλόμισθες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εμείς έχουμε ένα μισθό που μας επιτρέπει την συμφιλίωση. Εγώ έχω μια κόρη και ε, έναν άνδρα. Μπορώ βεβαίως ε, να πληρώσω και μια γυναίκα για να φροντίσει το, το παιδί μου. και προσπαθώ βεβαίως να είμαι ε, μαζί με το παιδί μου, αλλά μπορώ να πληρώσω και κάποιον άνθρωπο για να συμφιλιώσω την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, ενώ μια χαμηλόμιστη γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα, πολλές γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Λούλη, οι ίδιες για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να προωθήσουν ορισμένα πράγματα. Εγώ πριν να έχω παιδί σκεφτόμουν όπως λέγαν και άλλες γυναίκες ότι πρέπει να, είσαι, να συμπεριφέρεσαι κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά υπάρχουν ε, στοιχεία αστάθμητα Δηλαδή πολλές φορές πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο, να ακολουθείς ένα φρενιτιώδη ρυθμό. Και πολλές φορές τα παιδιά μας στην Ισπανία λένε προτιμώ να είμαι με τη γιαγιά και όχι με τη μαμά γιατί η μαμά είναι νευρωτική, είναι ιστερική. Δεν τη θέλω, προτιμώ τη γιαγιά που είναι ήσυχη. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε και την εκπαίδευση και τον τρόπο αντιμετώπισης να εργαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα στερεότυπα πραγματικά. Ε, η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέβομαι πλήρως αυτό το οποίο επισήμανε η προηγούμενη ομιλήτρια. Αυτό το οποίο νομίζω πως θα πρέπει να αποτελεί στόχο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο εθνικό επίπεδο είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να έχουν επιλογή οι γυναίκες αλλά θα πρέπει να μην φτάσουμε στην, ίδια στην οτροπία ότι οι γυναίκες είναι ίδιες με τους άντρες. Δεν θέμε να γίνουν οι γυναίκες ανθρακορίχοι. Γιατί να θέμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, μπορεί κάποιες γυναίκες να θέλουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα, αλλά ε, δεν νομίζω κανείς να τους αποτρέπει από το να κάνουν κάτι τέτοια, γιατί θυμάμαι στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία όταν έκαναν το ίδιο άντρες και γυναίκες με τα πενταετή σχέδια, κεντρικά διευθυνόμενη οικονομία. Ε, πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό. Αυτό, όπως λέει και η συνάδελφος, είναι η ομορφιά της ζωή. Θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να είναι και μητέρες οι γυναίκες και πρέπει να γνωρίζουμε το ότι το να είναι κανείς μητέρα είναι μια μεγάλη αξία και επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας. Και η φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να θεωρείται δουλειά, αμοιβόμενη. Γι' αυτό χαίρομαι για την υιοθέτηση της ε, οδηγίας ε, με την πρώτη ανάγνωση την περασμένη εβδομάδα στο Ρασβούργο. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις γυναίκες να σκέφτονται με τον τρόπο των ανδρών. Αυτό είναι και παραφύσιν. Ήμουν ε, εγώ διευθύντρια μεγάλου νοσοκομείου, έχω περάσει από διευθυντικές θέσεις αλλά ταυτόχρονα ήμουν τόσο χαρούμενη να ε, ε, κάτσω δύο χρόνια με το μωρό μου σπίτι, γιατί έχει και αυτό την αξία του και υπάρχει κάποια στιγμή ε, στην οποία πρέπει να προηγηθεί το μωρό και το παιδί. Βεβαίω, αυτό το οποίο συναντάω καμία φορά σε αυτήν εδώ μέσα την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι πως καμία φορά εστιάζουμε πάρα πολύ στα δικαιώματα των γυναικών εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών. Ε, εκεί πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Αυτό λείπει μέχρι στιγμής. Ε, με συγχωρείτε αν είμαι έτσι πολύ ειλικρινής. Σας ε, ευχαριστώ. Κυρία Κράτσα. εγώ θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια επενθύμηση ότι σήμερα με την δημόσια αυτή ακρόαση δεν θέτουμε επιτάπητος όλα τα προβλήματα της συμφιλίωσης και της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να τα πούμε, τα έχουμε ήδη πει και θα τα ξαναπούμε. Ε, συζητούμε για τις γυναίκες οι οποίες μπορούν να είναι σε ένα, μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά λόγω έλλειψης ορατότητας, έλλειψης βούλησης δεν είναι και έτσι πιστεύουμε ότι χάνει και η οικονομία και η κοινωνία και η επιχείρηση. Ήθελα να ζητήσω την κυρία Στάρας έτσι πολύ παραστατικά μας είπε τα προβλήματα της σύγχρονης ε, γυναίκας και μητέρας και τη συμμερίζομαι. Τι γίνεται με τον νόμο που υιοθετήθηκε στην Ισπανία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Έχει δοθεί μια περίοδος χάριτος από ό,τι ξέρω μέχρι να εφαρμοστεί με τις συνέπειες και τις κυρώσεις για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Ποια είναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ε, πληροφόρησή μας σήμερα να δούμε την εμπειρία της Ισπανίας μια χώρας η οποία υιοθέτησε από ό,τι ξέρω ένα νόμο αλλά θα τον εφαρμόσω από το 2015. Θα ήταν σημαντικό αν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση, πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις. Έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν κάτι. Ε, άρα αποδίδει η προοπτική μιας νομοθεσίας ή πρέπει αύριο να εφαρμοστεί μια νομοθεσία υποχρεωτικά, αλλιώ δεν κινείται τίποτα. Είναι κομβικό σημείο αυτό για μας. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κράτσα. Τώρα θα ήθελα να στραφώ προς τα μέλη του πάνελ έτσι ώστε εντάχει να μας σχολιάσουν εν είδη συμπεράσματος. Πέντε λεπτά, πέντε λεπτά η καθεμία. Η κυρία Σαμάν, Νατιβιντάντ και με την κυρία Πέναμ. Ναι, νομίζω πως η συζήτηση δεν ξέρω, ξεπέρασε ίσως το ζήτημα της ημερήσιας διάταξης. Να πω κάποια πράγματα για τη συζήτηση πρώτα. Μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση για τις εργαζόμενες γυναίκες ε, και την, ε, το εάν δικαιούται να δουλεύει με ίσους όρους με τον άντρα. Νόμιζα πως είχε τελειώσει αυτή η συζήτηση, οπότε θα την θεωρήσω λήξασα. Και από εκεί και πέρα. Για να φτάσουμε ξανά στην δυνατότητα των γυναικών να εξελιχθεί και να έχει τις ίδιες ε, δυνατότητες με τους άντρες. Θα ήθελα να πω πως δεν ήμουν η μόνη που το είπα. Μου άρεσε η προσέγγιση που ήταν και ποσόστοση που συνοδεύονταν με άλλα μέτρα που είχαν ξεκινήσει έτσι ώστε τα κορίτσια εξ αρχής να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα αγόρια και οι μητέρες να μπορούν να μοιραστούν τα καθήκοντα της οικογένειας όχι μόνο με την κοινωνία αλλά και με τους άντρες. Και οι άντρες ε, να θεωρούνται εξίσου με τις μητέρες για την οικογένεια και άλλα μέτρα με την πολιτική πίεση και τις εταιρείε και στον παρα... Το να μιλάμε για στερεότυπα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα για το ΔΣ είναι επίσης σημαντικό και θετικό είναι αυτό το οποίο ακούστηκε. Ε, ε, Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, ε, σημασία έχει η εκπαίδευση, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει εν μία νυχτή. Επίσης ακούστηκε πως κανείς δεν ανέφερε το θέμα της εκπαίδευσης των ανδρών στο ΔΣ. Είναι επειδή τώρα οι γυναίκες συζητάνε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που ανακύπτει το ζήτημα ε, αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε στην συζήτηση για το γιατί χρειάζεται να είναι κανείς σε ένα ΔΣ, τι απαιτείται και ίσως ρά αυτή των ικανοτήτων είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε, δηλαδή να δούμε πως θα εξετάζονται τα ζητήματα από διαφορετικές σκοπιές. Αλλά συμφωνώ, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα, πως εάν θέλουμε να πάμε στις ποσοστώσεις, θα πρέπει να συνοδευτούν από μέτρα. Δηλαδή μια βάση δεδομένων για να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες γενικές υποψήφιες. και να βρεθούν τρόποι παρακολούθησης και μέτρησης και πώς θα γίνουν απαραίτητες προσαρμογές αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στην Ισπανία, εγώ προέρχομαι από λατινική χώρα Ξέρω πως χρειάζεται κάποια παρακολούθηση για να φροντίσουμε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Θέλουμε το νόμο ή όχι. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς. Η κυρία Νατιβιτάντ. Ευχαριστώ. Ε, εμένα με λένε τη βασίλισσα των ποσοστώσεων. Γιατί θεωρώ πως κάτι γίνεται στην Ευρώπη, παίζει ηγετικό ρόλο και θέλω να αντικρούσω αυτό το οποίο ακούστηκε πριν, πως δεν συμβαίνει τίποτα. Χώρα-χώρα, ποσόστοση με την ποσόστοση, νόμο με τον νόμο, κάνετε αλλαγές, ανεξαρτήτως ο ένας από τον άλλον, που θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες που ελπίζω να είναι θετικές. Σε κανένα δεν αρέξει λέξη ποσόστοση, ούτε οι εταιρείε που θα το υποστούν, ούτε οι γυναίκες που θα επωφεληθούν. Ανακύπτει ένα ζήτημα και θέλω να αφαιρθώ εδώ πέρα στην Ιταλίδα στην Άλφο, της αξίας έναντι της ποσότητας. Δηλαδή ποσότητα έναντι ποιότητας. Και όταν μου το λέει αυτό μια γυναίκα, εγώ θέλω, μου λέει, να μπω στο σου επειδή είμαι φοβερή, όχι λόγω της ποσότητας. Και λέω ξεκόλα. Το ζήτημα είναι να μπει αυτή τη στιγμή μπει, ούτω ή άλλω θα πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει και πάλι θα απορριφθεί αν δεν τα κάνει. Η ποσόστοση είναι ένα τρόπο να μπούμε μέσα για να επιτύχουμε την ισότητα αμέσω. Παλεύουμε, έχουμε θετικές διακρίσεις της ΕΠΑ που επιτρέπουν στις γυναίκες να φτάσουν στις μέσες θέσεις διοίκησης και εκεί πέρα κολλάνε. Έχουμε την πλειοψηφία διευθυντών αλλά είμαστε μόνο 3% των διευθυνουσών συμβούλων και 16% της ανώτατης δίκης. Έχω βαρεθεί λοιπόν τους στόχους, το είπα και πριν. Οι ποσοστώσεις, εάν τις δείτε ως ένα μηχανισμό που ελπίζουμε θα είναι προσωρινός, μπορούν να μεταμορφώσουν την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι άντρες μας έφεραν σε αυτή την οικονομική κρίση. Ίσως λοιπόν οι γυναίκες μπορούν να διακυβερνήσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο είπατε πως συμφέρει τις επιχειρήσεις πρέπει να το δείτε στην Κομισιόν. Έχετε τόση έρευνα ήδη. Δηλαδή έχει ήδη υποθεί αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι οι άντρες θα προσκληθούν στην ακρόαση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Σωστό αυτό, αλλά πρέπει να προσέξετε ποιους Διευθύνονται σύμβουλου θα καλέσετε. Θέλετε αυτούς οι οποίοι πάνε καλά, αυτούς οι οποίοι δεν πάνε τόσο καλά και αυτούς οι οποίοι μπορούν να επηρεαστούν για να τα πάνε καλύτερα. Οι περισσότερες εταιρείε θα αντιπαλέψουν το να τους επιβάλλεται πράγματα. Έχουν υπάρξει αλλαγέ λόγω των ποσοστώσεων. Στη Γαλλία είχαν κολλήσει στο 7% οι γυναίκες στα Σίγμα. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση για τις ποσοστώσεις έφτασε το 14,4% μέσα σε τρία χρόνια. Μόνο και μόνο επειδή το συζητάνε. Δηλαδή έρχεται στο προσκήνιο με τρόπο που είναι μοναδικός. Να κάνει η Κομισιόν αυτό τον διάλογο με τους διευθύνοντες ε, συμβούλους και να καλέσει τον τύπο. Τα ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο εκπαίδευσης, έχετε απολύτως δίκιο, κάποιος το είπε, πως πρέπει να εκπαιδευτούν οι άντρες για την αξία. Την αξία στη σούμα, στον ισολογισμό. Να σας πω λοιπόν πως ήδη κάνετε αλλαγές και εσείς θα επιφέρετε αλλαγές σε άλλες χώρες. Η Νορβηγία έχει επενδύσει στις ΗΠΑ, έχουν επενδυτικά ταμεία και στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα της Παγκόσμια Τράπεζας ήταν η Νορβηγία θα ζητήσει από τις Αμερικανικές εταιρείε τις οποίες έχουν επενδύσει να αλλάξουν τα διοικητικά του συμβουλία. Πολύ μου άρεσε αυτή η ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νατιβιντάτ. Η κυρία Μπένα με έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ότι συμφωνώ με τη συνάδελφο γιατί ε, η χρηματοπιστωτική κρίση μας οδηγεί σε ένα άλλο τρόπο σκέψης. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί στην εκπαίδευση των γυναικών χωρίς να μιλήσουμε και χωρί, αν δεν δούμε αυτά τα, αυτό το μεγάλο ταλέντο που εκπροσωπούν οι γυναίκες, τότε δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να καταπολεμήσουμε ούτε την κρίση. Βεβαίως η ποσόστοση δεν είναι ευτυχής λέξη, αλλά είναι ένα προσωρινό ειδικό μέτρο εκκίνησης αυτής της διαδικασίας, αυτής της πρωτοβουλίας. Τη στιγμή που έχουμε τις γυναίκες εντός σε διευθυντικές θέσεις, τότε η αξιοκρατία θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Αλλά θα πρέπει να μπουν οι γυναίκες και αυτό το συζητάμε επί μακρόν. Γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε ο χρόνος για πραγματική δράση έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσει. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Κράτσα, έτσι ώστε να φτάσει σε ορισμένα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ και εσά που διευθύνατε αυτή τη συζήτηση και τις προσκεκλημένες μας που έδωσαν το δικό τους στίγμα, την εμπειρία τους τον ενθουσιασμό τους. Ε, μπορώ να σας πω ότι είναι από τις καλύτερες δημόσια ακροάσεις που κάναμε, γιατί ήταν όλες οι συγγήτριες πολύ συγκεκριμένες και πολύ ε, εστιασμένες στην ουσία του προβλήματος και των στόχων μας. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να μοιραστούμε κάποια συμπεράσματα, ότι το πρόβλημα είναι γενικό, δεν έχει ξεφύγει καμία χώρα από αυτό ε, και ότι τα αποτελέσματα στατιστικά είναι ενθαρρυντικά εκεί που υπήρξαν νομοθετικές και υποχρεωτικές παρεμβάσεις. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει αυτό, αποτελεί μια πραγματικότητα. Απορρίπτω και εγώ το δίλημα ποιότητα ή ποσότητα. Μπορούν να πηγαίνουν μαζί το ποιότητα ή ποσότητα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι στην Ιταλία επειδή είναι 3% η συμμετοχή των γυναικών στα υψηλά επίπεδα των, ε, συμβουλίων των εταιριών, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ικανές Ιταλίδες για να γίνει το 3, 8, 15, 20 και 40. Άρα σημαίνει ότι το θέμα δεν απασχολεί κανέναν και δύο πράγματα έχουμε μπροστά μας. Ή το αποδεχόμαστε ε, ή ε, λέμε ότι θα δράσουμε. Τώρα πώς θα δράσουμε. Εμείς, ξέρετε, το λέω και για τις φίλες μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην Ευρώπη ανταλλάσσουμε τις καλές πρακτικές μας, θέτουμε στόχους πολιτικούς να πάμε όλοι μαζί, αλλά ανακαλύπτουμε ότι στην πράξη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πάντα με τα ίδια βήματα, γιατί είμαστε σε πολλούς τομείς διαφορετικές πραγματικότητες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι έτοιμες να κάνουν ένα βήμα μπρος, υπάρχει μια οριμότητα. Γι' αυτό θα ήθελα την κυρία Στάρας, αν δεν μπορεί σήμερα κάποια άλλη φορά, να μας πει για την ισπανική εμπειρία, να δούμε αν η Ισπανία προετοιμάστηκε για αυτή την πραγματικότητα ή ήταν βία αποφασίστηκε ένας νόμος. Ε, από την άλλη πλευρά, πέρα από την οριμότητα, την παράδοση, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, υπάρχει το μέγεθος των εταιριών, ε, η παράδοση εταιρικής διακυβέρνησης και το διαφορετικό εταιρικό δίκαιο όπως είπε η κυρία Λούλινγκ. Λοιπόν, σίγουρα εμείς έχουμε να πάρουμε κάποιες παραμέτρους υπόψη, μας στην Ευρώπη, που, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ε, έχει ανάγκη να τις πάρει ε, μια άλλη χώρα μεγάλη, μικρή στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονό. Πέρασμα ότι πρέπει να δράσουμε. Από μόνο του το θέμα δεν προχωρεί, δεν προχώρησε πουθενά. Δεύτερον, ε, ο τρόπος της δράσης μας θα είναι περιθώρια διαβούλευσης, ε, ανάδειξη του προβλήματος, ε, θα δώσουμε εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς εταίρους ώστε θα προχωρήσουν σε ένα στάδιο μόνοι τους, θα, ζητήσουν, θα κάνουμε χρονοδιάγραμμα για την ομοθεσία, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι για να πετύχει αυτό το μέτρο, όπως για όλα τα μέτρα τα... που έχουν να κάνουν με ποσοστώσεις, πρέπει να συνοδεύεται από ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης πώ θα προετοιμαστούν οι γυναίκε για να παίξουν αυτό το ρόλο, πώ θα προετοιμαστεί η επιχείρηση για να δεχτεί αυτή την ε, αλλαγή, ε, η εκπαίδευση, ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, πώς, πώς εφαρμόζεται. Ε, δεν μπορεί, όταν εγκαταληφθεί ένα σχέδιο, έτσι μόνο του θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε αχ υποχρεωτικά να βάλω κάποιες γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τις βρω από την ιεραρχία της επιχείρησης, ψάχνω γυναίκες διάσημες από εδώ και από εκεί. Το βλέπουμε το ίδιο και στην πολιτική, ε, όπου δεν υπάρχει ένα, ένα συνοδευτικό σχέδιο για την ανάδειξη γυναικών ε, μέσα στα πολιτικά κόμματα, στην κοινωνία. Τρέχουν τελευταία στιγμή οι συνδυασμοί να βρουν γυναίκες για να κάνουν το καθήκον τους προς την ομοθεσία. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε προ μιας πολύπλευρης πρόκλησης στην οποία θα, θα ανταποκριθούμε, πιστεύω, και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βελγική Προεδρία και η Ουγγρική αργότερα. Ε, το θέμα είναι ότι μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις ε, ανησυχίες και αυτές τους στόχους ε, με ε, γυναίκες που, που εκφράζουν, όπως το είδαμε σήμερα, φορείς που αγωνίζονται για αυτό, το, αυτή την υπόθεση τόσο στην Ευρώπη όσο και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, όσο και σε global επίπεδο που είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό. Αυτά ήθελα να πω, ε, κυρία Πρόεδρε, σαν γενικά μέτρα, σαν γενικά συμπεράσματα και πάλι να ευχαριστήσω και εσάς, τις συνομιλήτρες και τα μέλη μας που έμειναν μέχρι αργά να συζητήσουν και να ακούσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κράτα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που αναλάβατε την πρωτοβουλία να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σήμερα η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή και ζωντανή και μας επέτρεψε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει. Ευχαριστώ όλες τις ομιλήτριες του πάνελ και εσάς που το οργανώσατε. Οι ομιλήτριες συνεισέφεραν πολύ θετικά στη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσία της και την άποψή της και, τις, και τους συναδέλφους που παρέμειναν μέχρι το τέλος. Η συζήτηση νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη. Καμιά φορά ακούστηκαν και διαφωνιούλες, αλλά καλό είναι πάντοτε να υπάρχει συζήτηση για να ακούγονται όλες οι απόψεις και να, βρίσκεται, να βρίσκουμε έτσι τον καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε. Είμαι πεπισμένη στην έκθεσή της η κυρία Κράτσα θα βρει αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ επίσης τη γραμματεία που εργάστηκε τόσο σκληρά για τη διοργάνωση της ακρόασης αυτής και βεβαίως και τις εξαιρετικές διερμηνεύτριές μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και θα ξαναβρεθούμε αύριο στις 9.